Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, καθίστε για να αρχίσουμε. Διότι έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη, έχουμε και συνάντηση συντονιστών και ψηφοφορία στις 11. Άρα πρέπει να αρχίσουμε τώρα και να έχουμε την ώρα υπόψη μας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να ανακοινώσω. Το σημείο 4 για την προστασία του ευρώ κατά της παραχάραξης η εισηγήτρια η κυρία Μάκεντάιρ ζητεί να αναβληθεί μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Τα σημεία 5 και 12 έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ τους. Η έκθεση Κέρκοπ για τα ευρωπαϊκά στατιστικά για την ασφάλεια από το έγκλημα θα αρχίσει 9 και 25 σήμερα και η παρουσίαση από τον διευθυντή της Frontex Ilka Λάιτινεν θα λάβει χώρα στις 11 και 20. Επίσης, οι ψηφοφορίες θα αναβληθούν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ η επόμενη συνεδρίαση είναι 5-6 Νοεμβρίου. Είναι το σχέδιο έκθεσης για το πολιετές ε, πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, έκθεση της Ντανόκα. Ε, σχέδιο έκθεσης για την κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2012-2011. Η συγγήτρια είναι η κυρία Φλαζίκο Βαμπένοβα εδώ και ο κύριος Κοέλιο θα λάβει το λόγο για να ενημερώσει την Επιτροπή για τη το πέρασμα στη OSIS δεύτερης γενιάς, το 2. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Και πάμε στο σημείο 2, που είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου. Καλωσορίζομαι τον κύριο Νταβίδ Σασόλη που έγινε ε, αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή μας αντί για την κυρία Καταρίνα Νεβεντάλοβα. Επίσης ανακοινώνω ορισμό εισηγητών όπως συμφωνήθηκε από τους συντονιστές στη συνεδρίασή τους. Την κυρία, όχι, τον κύριο, συγγνώμη, τον κύριο Μαριάν Ζων Μαρινέσκου, που είναι εισηγητής για την έκθεση Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων. Ο κύριος Κλοντ Μωράης ε, είναι εισηγητής στην έκθεση Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για τη διευκόλυνση των εκδόσεων θεωρήσεων. Και εγώ ο ίδιος ε, έχω οριστεί εισηγητής, ε, ορίστηκα εισηγητής για την έκθεση με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης ε, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ε, μέσω του ποινικού δικαίου. Και υπάρχει και μια, ένας ορισμός ε, συντακτών γνωμοδοτήσεων, ο κύριος Πέτρο Κωνσταντίν Λουάν για τη γνωμοδότηση, βασικά έγγραφα πληροφόρησης για προϊόντα επενδυτικά. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Στα... Α, στο τρίτο σημείο έγκριση των πρακτικών βλέπω, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Και πάμε στο πρώτο θέμα ουσία, στο σημείο 4, που είχε συμπεριληφθεί ε, στην ε, ημερήσια διάταξη. Αυτό όμως αναβάλλεται, είναι η έκθεση McIntyre και περνάμε κατευθείαν στις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με την ασφάλεια από την εγκληματικότητα. Ο κύριος Κίρκοπ είναι... Α, εκπροσωπείται από τον κύριο Άσουερθ από ό,τι κατάλαβα. Εμείς θα δούμε το σχέδιο έκθεσης που επεξεργάστηκε ο κύριος Κίρκοπ για την πρόταση που έχει συζητηθεί ήδη στην Επιτροπή εντατικά με τους σκιώδεις εισηγητές. Υπάρχουν θέματα που αφορούν τη μεθοδολογία και το κόστος της πρότασης. Ο κύριος Άσουερθ θα μας μιλήσει ε, εξ ονόματος του κυρίου Κέρκοπ και μετά θα θέσω με προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Κύριε Άσουερθ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώνω ότι ο κύριος Κέρκοπ δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει εδώ. Ο συνάδελφος Άνθεα Μάκινταρ θα παρουσίαζε την έκθεση, αλλά πρέπει να σας αναφέρω ότι το προηγούμενο διήμερο ε, ε, σε ένα τύχημα έσπασε το πόδι της και θα μείνει για κάποιο διάστημα μακράν του Κοινοβουλίου. Συμφώνησα λοιπόν να διαβάσω το σύντομο, τη σύντομη ανακοίνωση του κυρίου Κέρκοπ. Παραθέτω από την έκθεσή του Λέει ότι χαιρετίζει την ευκαιρία για μια ακόμα ανταλλαγή απόψεων πριν από την ψηφοφορία στην Επιτροπή για να εκφράσει την άποψή του ως εισηγητής για τους άλλους ε, ε εισηγητές που θα παρουσιάσουν απόψεις και να παρουσιάσει την επεξηγηματική έκθεση που ζητεί απόρριψη αυτής της πρότασης. Μετά από διεξοδικές συζητήσεις ε, με άλλους συζητητές και μετά την συνάντηση με την Κομισιόν και τη Eurostat πολλές φορές και ε, μετά από μια συνάντηση μεταξύ Eurostat και άλλων σκιωδών εισηγητών κατέστη σαφές ότι ως νομοθέτες δεν βλέπουμε επαρκή προστιθέμενη αξία που να δικαιολογεί τη συνέχιση της πρότασης αυτής. Το, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αναφέρει και παραθέτω εδώ ε, επαρκή, αξιόπιστα, συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία που είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για ε, την ανάγκη ανάληψης δράσης, ε, για την εφαρμογή αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Τέλος του παραθέματος. Συμφωνώ ότι τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν καλή βάση για να ξέρουμε πώς θα στοχεύσουμε στην μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία και θα πρέπει να κάνουμε εκθέσεις, να διώκουμε ε, το έγκλημα και να υποβάλουμε αναφορές για αυτά. Με τα 12 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό, ο εισηγητής λέει ότι παραμένει πεπισμένος σε σχέση με την προϊωστηθέμενη αξία αυτής της μορφής ερευνών και των δεδομένων που θα είναι αμφισβητήσιμα. Σχετικά με τη μεθοδολογία ε, όμως παραμένουν κάποια ερωτηματικά ε, γιατί ε, υπάρχει θέμα ειλικρίνειας απαντήσεων και έτσι δεν συνάγεται προς τη θέμενη αξία. Μπορεί να υπάρξουν και παρερμηνίες. Η υποκειμετικότητα και η ε, και τα, τα ευαίσθητα θέματα που πολλές φορές ε, τίθενται μέσα από τους τύπους των ερωτήσεων προκαλούν ε, άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση του ερωτώμενου σε προβλήματα ναρκωτικών ή την ιδιοκτησία όπλων ή το φόβο της τρομοκρατίας. Είναι δύσκολο να δούμε ότι η αξία που θα βγάλουμε σχετικά με τη είναι, είναι δύσκολο να συναγάγουμε στατιστικά στοιχεία. Ε, είναι διαφορετική η αντίληψη που έχει κάποιος για τα εγκλήματα αυτά. Μία δαπανηρή ε, έρευνα χωρίς να δώσει τα απαραίτητα αποτελέσματα θα ήταν ανεύθυνη. Ο εισηγητής λέει ότι υπογραμμίζει ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο του Eurostat και το, την αξία που μπορούν να έχουν τα στατιστικά στοιχεία. Προτείνει όμως ο εισηγητής να απορρίψει την πρόταση η Επιτροπή. Τα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν ε, σε σχέση με το διασυνοριακό έγκλημα σε όλες τις μορφές του, είτε είναι... Ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών ανθρώπων, ε, κυβερνοέγκλημα, λέει ότι θα ενθάρρυνε την Κομισιόν αντίθετα να υποβάλει μια εναλλακτική πρόταση η οποία θα στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όπου θα υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με την ε, σχέση κόστους ωφέλους αλλά και την προστιθέμενη αξία του εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο, ο κύριος Ντεγιόν, η κυρία Ντέλεγαντ, κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή μας κύριο Κέρκοπ. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ γενναίο να ε, εμένει στην πρόταση απόρριψης της πρότασης της Κομισιόν, όμως είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση ε, ε, στη δεδομένη περίπτωση. Πήραμε και μία επιστολή από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δεν ε, αναφέρεται στις αντιρρήσεις μας. Λέει όμως ότι αυτές οι στατιστικές είναι πολύτιμες. Βεβαίως, εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι. Εμείς είπαμε τρία πράγματα επιχειρηματολογώντας και δεν θα μακρηγορήσω γιατί ε, ε συμφωνώ με τον εισηγητή. Πρώτον πρέπει να ε, δούμε χρειάζονται αυτά τα δεδομένα. Χρειάζονται κατά προτεραιότητα ε, σε σχέση με δεδομένα για παράδειγμα για το διασυνοριακό έγκλημα που είναι πιο μεγάλη προτεραιότητα ε, από το εθνικό έγκλημα και βέβαια στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών μπορεί να θέλει κανείς να ανταλλάσσει δεδομένα και για εθνικά εγκλήματα δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Δεύτερον η Κομισιόν θα πρέπει να ρυθμίσει ε, εν πάση λεπτομερία όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια τέτοια μελέτη σε ευρωπαϊκή κλίμακα ή μπορούμε εδώ να επαφιέμεθα στις εθνικές υπηρεσίες. Και πριν συμφωνήσω σε μια τέτοια πρόταση θα ήθελα να κάνω ένα γύρο τραπεζιού με τις εθνικές υπηρεσίες και να μας πούν γιατί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, γιατί έτσι περνώ στο τρίτο επιχείρημά μου. Εάν ανταποκριθούν και δώσουν τα παραδοτέα, και σε πολλές χώρες υπάρχουν στοιχεία τέτοια μακροδεδομένα που θέλει να πάρει η Κομισιόν, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ε, που θα μας βοηθήσουν σε θέματα ποιότητας και πώς θα οργανωθούν, γιατί έχουν εμπειρία, τα κάνουν όλα αυτά εδώ και πολύ καιρό. Και μετά θα έχουμε ένα μηχανισμό κόστους αποτελεσματικότητας ε, που θα δουλεύει ε, καλά, δεν θα κάνει επικαλύψεις και θα έχει μια έξυπνη μεθοδολογία. Πολλές ε, φορές μιλήσαμε για τις ε, προτάσεις αυτές της Κομισιόν. Δεν θα τα ξαναπούμε γιατί δεν έχει είναι και αστείο να τα πούμε τρεις φορές. Αλλά όταν ρωτάμε κάποιον πώς αισθάνεται ή να τον ρωτήσουμε αν οπλοφορεί, μα πώς θα πάρουμε από αυτά, από αυτές τις υποκειμενικές ερωτήσεις αντικειμενικά στοιχεία. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας κατά με ότι η προετοιμασία της Κομισιόν δεν είναι η πρέπουσα και συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Κέρκο ότι πρέπει να την αποσύρει η Κομισιόν. Μην χάνουμε χρόνο, μην δίνουμε πόρους σε αυτό το θέμα, να την πάρει πίσω ως ενήλικοι να δεχτούν, να, να παραδεχτούν ότι δεν έγινε σωστά η δουλειά και πρέπει να ξαναγίνει. Κυρία Σδανόκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Ούλρη και Λούνατσεκ που είναι σκιώδης εισηγήτρια και εκπροσωπεί τις απόψεις των πρασίμων. Και εγώ. πρέπει να προσέξουμε όταν έχουμε τέτοιες δαπανηρές προτάσεις, ιδιαίτερα δεδομένες της σημερινής οικονομικής κατάστασης. Πρέπει να καταδειχθεί σημαντική προστιθέμενη αξία για να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση. Πιστεύουμε ότι είναι δύσκολο να συγκρίνουμε στατιστικά στοιχεία στο έγκλημα, εκτός και αν έχουμε πλήρως εναρμονισμένο ποινικό δίκαιο. Και εδώ δεν συμφωνούμε. Πρέπει να ελέγξουμε αν η Κομισιόν είναι ο αρμόδιος φορέας για να συντονίζει τα στατιστικά στοιχεία. Ίσως ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να είναι καλύτερος. Τέλος, πολύ σημαντικό, θα πρέπει να δούμε τι, τα προβλήματα που θέτει και το EDPS. Μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν με την πρόταση απόρριψης που υποβάλλει ο κύριος Κέρκοπ. Με μία επιφύλαξη όμως. Δεν είμαστε κατά της ιδέας καταρχήν, αλλά η πρόταση θα πρέπει να είναι λιγότερο δαπανηρή και πιο ορθή. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζίλστερ, ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την έκθεση του κυρίου Κίρκοπ. Αναρωτιέμαι μάλιστα στο συμφέρον που έχει η Κομισιόν να συλλέξει τα στοιχεία αυτά. Στην ε, Πολωνία, μία έρευνα της αστυνομίας διεπ διαπίστωσε ότι η εγκληματικότητα ε, έχει μειωθεί, διότι έχει μεταφερθεί σε άλλες χώρες. Η έρευνα αυτή διαπιστώνει ότι τελικά η Πολωνία ε, ε, εξάγει βία. Είναι δυστυχές, αλλά δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Επίσης, σχετικά με τη διασυνοριακή εγκληματικότητα, έχουμε υποβάλει ερωτήματα στο Συμβούλιο ε, και κάθε φορά η απάντηση είναι η ίδια, δέστε τα στοιχεία στην Eurostat. Ε, όμως τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αφορούν το έτος 2008, επομένως δεν είναι επικαιροποιημένα. Τώρα, στην στατιστική βλέπουμε την ε, εξέλιξη αναχώρα και ανα ε, έγκλημα, αλλά δεν έχουμε όμως ε, στοιχεία για την διασυνοριακή εγκληματικότητα. Επομένως ερώτημα, Οι Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν έχουν γνώση των συγκεκριμένων στοιχείων που συλλέγει η Eurostat και το Κοινοβούλιο από τη δικιά του την πλευρά δεν ε, μπορεί να αρκεστεί στα στοιχεία ε, της, ε, της στατιστικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και συγκρίσιμα. Εδώ όμως βλέπουμε ότι είναι απαρχιωμένα, ότι δεν υπάρχει καμία προστιθέμενη αξία στα στατιστικά αυτά στοιχεία. Δεν έχουμε καμία αναφορά στο διασυνοριακή εγκληματικότητα κτλ. Επομένως για να μπορέσουμε να έχουμε σωστά στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία. Επομένως, στηρίζω τον εισηγητή, η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη τη σοβαρά το θέμα αυτό και να ε, έχει πάντα γνώμονα την, ε, τον ρεαλισμό και την πραγματικότητα. Έχουμε πολλές ε, παρεμβάσεις. Ο κύριος Μπουζούτιλ, ναι σας έχω δει κύριε Μπουζούτιλ. Θέλετε να μιλήσετε τώρα. Ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία, μόλις έφτασα. Η θέση του ΕΛΚΑ είναι να ακολουθήσουμε την ε, πρόταση του εισηγητή. Δεν είμαστε ακόμα πεπισμένοι <clears throat> απολύτως για τον ε, λόγο ύπαρξης ε, της πρότασης αυτής. Μόλις έφτασα δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι αυτό, ότι ακολουθούμε την πρόταση του εισηγητού. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος, Ashworth. Θέλετε να αντιδράσετε σε κάποια σχόλια. δεν θα αντιδράσω, γιατί ο συνάδελφος κύριος ε, Κίρκοπ ε, είναι αυτός ο οποίος ε, έχει αναλάβει την έκθεση, αλλά βεβαίως εγώ θα του πω εν λεπτομερία τα όσα υπόθηκαν στην Επιτροπή μας και βεβαίως να πω ότι είμαι ευγνώμων για τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι. Η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο τώρα, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε την δυνατότητα να προσπαθήσουμε να, αποφέρουμε κάποιες, να επιφέρουμε κάποιες ερωτήσεις, α, απαντήσεις. Λέγομαι Εδωάδρο Ανδρέδο και είμαι υπεύθυνο για τις κοινωνικές στατιστικές της Eurostat. Νομίζω ότι δεν πρέπει, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να σας πείσουμε για την σημασία ύπαρξης ε, στατιστικών στοιχείων, ε, δεδομένων, ε, για να δούμε πώς λειτουργούν οι στατιστικές. Την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, είδαμε την έγκριση ενός νέου νόμου που θα βελτιώσει τη θέση των, των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών απανταχού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, και είναι απόρρια της οδηγίας για τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των θυμάτων. Επίσης ε, υπάρχουν ευάλωτοι ε, πληθυσμοί, ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που θέλουμε να προστατεύσουμε. Αλλά πόσοι είναι αυτοί οι πληθυσμοί, πόσα είναι τα θύματα, πώς κατανέμονται, έχουν αυξηθεί ή έχουν μειωθεί. Υπάρχουν κάποια ομάδε οι οποίε είναι περισσότερο εκτεθειμένε από άλλε επίση σε σχέση με, τους, ε, ε, με τι ομάδε αυτέ. Ε, τι γνωρίζουμε, έχουμε διοικητικά Μητρώα στρέφονται προς την αστυνομία ή προς άλλες αρχές. Τα θύματα αυτά έχουμε μητρώα για τις προσφυγές τους. Επομένως αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θέλουμε να απαντήσουμε και κάποιοι από τις βουλευτές είπαν ότι οι παρούσες πληροφορίες δεν είναι αρκετές, άρα χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία και συμφωνούμε με αυτό. Το κείμενο του κανονισμού που προτείνομαι ε, ε, δίνει απαντήσεις σε μια ε, πολύ σημαντική σειρά μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί βάση των συνθηκών της Χάγης ή της Στοκχόλμης. Θέλουμε να κάνουμε πολιτική βάση συγκεκριμένων στοιχείων, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν θέλω να πείσω κανέναν εδώ μέσα ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα που είναι εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Στατιστική στατιστική υπηρεσία και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες είναι το καλύτερο σώμα το οποίο θα καθορίσει τις αρχές συλλογής στατιστικών στοιχείων. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής ε, Στατιστικής Κοινότητας τελικά είναι ε, ε, ομού και σε συνεργασία αυτή η πρόταση. Το 2010 είχαμε το εγχειρίδιο για την θυματοποίηση ε, και, μας, και αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν βάση σε μια σειρά πολυερωτικών προγραμμάτων που ξεκίνησαν ήδη από το 2008 και το 2010 σε 16 χώρες μέλη και που προετοίμασαν το έδαφος για το κείμενο το οποίο έχετε τώρα μπροστά σας. Η ανάπτυξη αυτών των ε, ερευνών ε, έχει πάει πάρα πολύ καλά για την ώρα και μάλιστα κέρδισε το βραβείο της Στοχόλμης για την ε, για τις εγκληματικές έρευνες το 2012. Βεβαίως εμείς αναπτύσσουμε, έχουμε αναπτύξει ε, και ομάδες μελέτης και ομάδες εργασίας σε επίπεδο στατιστικής ε, κοινότητας και επομένως έχουμε προωθήσει κάποια από τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην οδηγία. Όσον αφορά την έρευνα για τη θυματοποίηση, έχουμε βασιστεί και στις, προτα... και στις αντίστοιχες έρευνες της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, βεβαίως κατανοούμε ότι το θέμα είναι σημαντικό και γύρονται πολλά ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι θα ξέρετε ότι ε, έχει ήδη συζητηθεί το ζήτημα στον το Συμβούλιο και έχουν υποβληθεί τροπολογίες οι οποίες <clears throat> εμπλουτίζουν το κείμενο. εκπλησόμεθα που δεν ε, ε, μπορεί να γίνει μια ανάλυση αντίστοιχη με αυτή που έγινε στο Συμβούλιο με την Επιτροπή σας εδώ. Γιατί και στο Συμβούλιο όταν δεν υπάρχει ομόφωνη θέση γίνεται, ε, λαμβάνονται αποφάσεις και γίνεται συζήτηση βάσει πλειοψηφιών. Νομίζουμε πάντως ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε στοιχεία και όσον αφορά ε, και την ε, θυματοποίηση και βεβαίως όλα τα στοιχεία ε, θα ληφθούν υπόψη και θα καταγραφούν στα διοικητικά μητρό τα οποία τώρα συστήνονται. Βεβαίως όλα τα στοιχεία θα είναι απόρριτα ε, και μην ξεχνούμε ότι σε πολλές χώρες μέλη προβλέπεται ποινή φυλάκισης για περιπτώσεις ε, παραβίασης ε, του στατιστικού απορρίτου. Πολύ σύντομα να απαντήσω σε κάποιες από τις επικρίσεις που αναφέρθηκαν αναφέρεται ότι το εργαλείο που προτείνονται δεν είναι συνεκτικά. Ε, εμείς ετοιμάζουμε κείμενο για την ε, εναρμονισμένη εφαρμογή. Κάποιες χώρες ε, θέλουν, προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους ερευνητικές τομές, δομές συγγνώμη, και εν πάση περιπτώσει το κείμενο προβλέπει αρκετή ευελιξία σε αυτό. Επίσης το θέμα της υποκειμενικότητας των απαντήσεων ή της δυνητικής υποκειμενικότητας των απαντήσεων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να απαντά ο ερωτώμενος στις ε, ερωτήσεις που του τίθενται και επομένως θα απαντήσει βάσει της προσωπικής του εκτίμησης εάν του ζητούμε την προσωπική του αντίληψη. Επίσης αμφισβητείται ε, βάσει της εκθέσεως ε, η εισαγωγή κάποιων παραμέτρων. Αλλά βεβαίως την έρευνα θα πρέπει κανείς να τη δει σαν ένα σύνολο. Πρόκειται για μια κοινωνικού περιεχομένου έρευνα. Υπάρχουν κάποιες μεταβλητές ε, οι οποίες εκτός περιεχομένου μπορεί να φαίνονται χωρίς ουσία και ανεφλόγου, όμως εάν τις δει κανείς σαν σύνολο είναι πάρα πολύ λογικές. Επίσης, ε, η δειγματοληψία είναι σημαντικό στοιχείο uh, It goes without saying, as I said ε, ε, επομένως η τυχεοποίηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην έρευνα και βεβαίως εμείς οπωσδήποτε θα δώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα δώσουμε και συνοπτικές παρουσιάσεις των πινάκων. Ε, μην λησμονείτε ότι όλες οι κοινωνικές στατιστικές, ε, Ευρώπη 20-20 δείκτες, ε, όλες οι στρατηγικές για την ανεργία, για τα κοινωνικά συστήματα βασίζονται στις κοινωνικού περιεχομένου έρευνες. Η έρευνα για την ένδια είναι αυτή η οποία οδήγησε στην τροποποίηση τριών δικτών. Επομένως, ναι, είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που ε, κάνουμε τέτοια έρευνα. Και ναι, συνηθίζονται τέτοιου είδους έρευνα. όσον αφορά τώρα το κόστος της άσκησης αυτής. Όπως σας είπα, ξεκινήσαμε πιλωτικά προγράμματα και έχουμε εν λεπτομερία ε, προδιαγράψει τα ε, ποσά και βεβαίως για να έχει κανείς, να επιτύχει κανείς καλά και ε, αξιόπιστα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, αντίστοιχα στάνταρ σε όλες τις αρχές. Έχουμε προβλέψει 12 εκατομμύρια για, την, για ένα εκατομμύριο ερωτόμενους και μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία της έρευνας φτάνουμε σε ένα ποσό Τη τάξη των 45 ευρώ ερωτώμενο που είναι ε, φυσιολογικό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την ε, ευρωπαϊκή στατιστική. Όταν οι καλύτεροι Ευρωπαίοι στατιστικολόγοι ε, συνδυάζουν τις προσπάθειές τους, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Ε, πιστεύουμε, είμαστε πεπισμένοι ότι η έρευνα αυτή θα δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε πολύ ουσιώδεις τομείς όπως είναι ας πούμε τα θύματα. Και στην ε, ε, οδηγία για το δημογραφικό βλέπουμε ότι υπάρχουν αιτήματα τα οποία σχετίζονται ε, με στατιστικές έρευνες. Επομένως αυτό είναι το εργαλείο το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας. Και σαν ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται για διαδικασίες που ξεκίνησαν στη Χάγη και στη Στοκχόλμη και τις συνεχίζουμε. Περαίνοντας να πω ότι λυπούμε στα ειλικρινά για την απόρριψη ε, της ε, πρότασης. Ε, λυπούμαστε για την θέση που παίρνει η Επιτροπή σας, αλλά βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Κομισιόν για την συμβολή αυτή. Κύριε Μπουσουτήλ, θέλετε να πείτε κάτι? δεν πρόβλημα. Ναι, πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Είναι κρίμα που είναι τόσο λίγοι συνάδελφοι παρόντες σήμερα το πρωί, γιατί είναι σημαντική η απόφαση απόρριψης μιας πρότασης της Κομισιόν πάντοτε. Άκουσα πολύ προσεκτικά την ε, παθιασμένη αυτή έκκληση του εκπροσώπου της Κομισιόν. Το ΕΛΚ είναι υπέρ της υποστήριξης του εισηγητή γιατί δεν βλέπουμε λόγο να ε, αλλάξουμε τα ευρήματα που μας παρουσιάζει ο εισηγητής. Αν όμως η Κομισιόν καταφέρει να πείσει τον εισηγητή να βρουν μια συμβιβαστική λύση στο θέμα αυτό, τότε και εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον εισηγητή, αν θέλει να αρχίσει με την Κομισιόν να ψάξει να βρει κάποιο τρόπο διεξόδου από το αδιέξοδο. Έχουμε κάποια λεπτά στη διάθεσή μας, ε, περιμένουμε την κυρία Βέμπερ που είναι υπεύθυνη συγγήτρια για το επόμενο θέμα, οπότε αν θέλετε να πείτε κύριε Ντεγιόν κάτι ακόμα, ευχαρίστω και ο κύριος Άσουορθ επίσης αν θέλει να κάνει τελικές παρατηρήσεις αφού ακούσατε την Κομισιόν ε, και τους δύο συναδέλφους που μίλησαν, ο κύριος Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όσον αφορά αυτά που είπε μόλις ο κύριος Μπουσούτιλ. Ε, όλα αυτά κοστίζουν χρήματα. Και εμείς κοστίζουμε χρήματα. Και βλέποντας ε, και πόσα πράγματα έχουμε στο τραπέζι στην ε, Επιτροπή μας, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ξοδέψουμε κι άλλο χρόνο σε, για να ξοδέψουμε πάνω σε μια κακή πρόταση έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να τα βολέψουμε για να βγούμε από το αδιέξοδο. Η Κομισιόν είναι αυτή η οποία πρέπει να βελτιώσει την πρότασή της. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ξαναμπούμε σε ε, ακόμα έναν ατέρμονα γύρω ανώφελων συζητήσεων. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο διασυνοριακό έγκλημα για το οποίο υπήρχε συγκεκριμένη εντολή και το οποίο συζητήσαμε επιμακρών ε, στην Επιτροπή μας έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε σωστά και το εθνικό ή τοπικό έγκλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. <clears throat> Δεν είναι απολύτως σαφές ότι χρειαζόμαστε ε, ομαδοποιημένα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, σε αυτό το έγγραφο της ε, Κομισιόν δεν εξηγείται καλά η πρόταση και δεν μας εξηγούν γιατί δεν μπορούμε καθόλου να βασιστούμε στα αστυνομικά αρχεία. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες δεν ε, έχουν αξιόπιστα στοιχεία και επομένως η πρώτη μου κίνηση θα ήταν να ε, βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτές τις συγκεκριμένε περιπτώσεις και σε αυτές τις συγκεκριμένε χώρε, έτσι ώστε τα αστυνομικά μητρώα να είναι, τα αστυνομικά αρχεία να είναι αξιόπιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να ξαναμπούμε σε αυτήν την ε, συζήτηση. Έχουμε εξηγήσει εν λεπτομερία γιατί θεωρούμε τη μεθοδολογία εσφαλμένη. Και τι να σας πω, εάν αυτό ε, ε, αγαπητέ εκπρόσωπο της Κομισιόν είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των υψηλού επίπεδου συναντήσεων που μας αναφέρατε, τότε λυπούμαστε. Μη μας κάνετε να χάσουμε κι άλλο χρόνο. Πάρτε πίσω την πρόταση, κάντε την καλύτερη, βελτιώστε την και τότε να μιλήσουμε. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δικές μου διαπιστώσεις δεν είναι διαφορετικές από αυτές τις, ε, από αυτές τις κομισιόν. Εμάς μας επαναπέμπουν τις ε, κριτικές. Το βασικό αίτημα είναι υπέρ της ε, ποιοτικής έρευνας κατά της ε, ποσοτικής. Βέβαια δεν πετάω τη σκούφια μου για την ποιότητα της πρότασης. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές ως προς τις πολιτιστικές συμβάσεις των ε, κρατών μελών. Αυτό όμως δεν εμποδίζει μια μεγάλη συγκρισιμότητα ε, και ανησυχώ και για τη θέση του ΕΛΚ που θέλει να υποκύψει στη νέα πρόταση της Κομισιόν. Η Προεδρία έχει κάτι να πει. Η Κυπριακή Προεδρία. Ε, εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η πρόταση κανονισμού για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με την ασφάλεια από την εγκληματικότητα συζητήθηκε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές κατά τη διάρκεια πέντε συναντήσεων ε, υπό Πολωνικής Προεδρίας, αρχής γενομένης στις 12 Ιουλίου 2011. Ε, ως αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων, η Πολωνική Προεδρία ετοίμασε στις 22 Δεκεμβρίου 2011 μια συμβιβαστική πρόταση. Όπως ανέφερε και η Επιτροπή, το Συμβούλιο προχώρησε σε τροπολογίες προκειμένου να βελτιώσει τη σχετική πρόταση. Ε, ορισμένα κράτη-μέλη έθεσαν ωστόσο γενική επιφύλαξη ως προς την πρόταση αυτή. Ε, να σημειώσω εδώ ότι η πρόταση αυτή δεν ε, έχει συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο, παρά μόνο σε επίπεδο ε, εμπειρογνωμόνων στην ομάδα εργασία. Η Κυπριακή Προεδρία θα περιμένει την τελική έκθεση τη Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ, προκειμένου να διαφανεί ο τρόπο χειρισμού του συγκεκριμένου φακέλου. Ευχαριστώ. Now back to you, Mr. Ashworth.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 Ε, θα μεταφέρω στον κύριο από όλα τα στοιχεία αυτά και ευχαριστώ πολύ ε, όλους τους συναδέλφους ε, που έκαναν σχόλια. Κυρίως θα αναφερθώ στα σχόλια που κάνατε στον εισηγητή και την δυνατότητα περαιτέρω συζητήσεως του όλου θέματος. Νομίζω ότι το θέμα εδώ είναι εάν το, εάν το θέμα αξίζει, το αποτέλεσμα αξίζει τα λεφτά του και εδώ μιλάω σαν μέλος της Επιτροπής προπολογισμών. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα και η προστιθέμενη αξία αξίζει ε, τα χρήματα τα οποία το κόστο που θα έχει αυτή η έρευνα. Επομένω, θα πρέπει να έχουμε πληροφορίε, τις οποίε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, <clears throat> με άλλο τρόπο, δηλαδή είτε από εθνικές στατιστικές είτε με ε, οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αλλά βεβαίως όλα αυτά τα στοιχεία θα τα δώσω στον κύριο Κίρκοπ άμα τη επιστροφή του και θα σας τα μεταφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Κίρκοβ για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο, όπως είπα και προηγουμένως, γιατί στις 11 έτσι κι αλλιώς έχουμε άλλη δουλειά. Η κυρία Βέμπερ. Η κυρία Βέμπερ έρχεται από ό,τι μου λένε. Λέω λοιπόν να καθίσουμε εδώ, μην κάνουμε διάλειμμα, γιατί θα χάσουμε χρόνο. Ας κάτσουμε εδώ, σε ένα λεπτό μου λένε ότι θα έρθει. Ευχαριστώ. yes, yes, yes, yes. Yes. Yes, excuse me. I, I forgot Συγγνώμη. Ξέχασα να πω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση Kirchhoff είναι η 16 Οκτωβρίου. Πέντε μέρες από τώρα, στις 17 ώρες. 5 το απόγευμα. Αυτή είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Σημειώστε την όσοι συμμετείχατε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Hello. Thank Καλώς ήρθατε κυρία Βέμπερ. Δεν κάναμε διάλειμμα. Είπαμε στους συναδέλφους ότι θα ερχόσαστε ανα πάσα στιγμή και να σας λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 6 που είναι ο, Ευρωπαϊκός, ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρότυπες ρυθμίσεις. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Είχε προγραμματιστεί για τις 10 η έκθεση και θα έπρεπε και το κέντρο για την ελευθερία των μέσων να έρθει εδώ να παρουσιάσει τις απόψεις τους και να συμμετέχουν. Και είναι επίσης καθοδόν. Δηλαδή τι λέτε να τους περιμένουμε. Κοιτάζω γύρω μου επίσης και δεν βλέπω και τους σκιώδεις. Α, α εσείς έχετε αναλάβει. Καλώς. Α, εντάξει. Ε, αντικαταστάσεις πολλές στους κοιόδης. Ο ε, δικός μου δεν είναι εδώ. Αν αναλαμβάνετε και καθ' ολοκληρία, εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνω την κατάσταση που διαμορφώθηκε, γιατί έπρεπε να αναδιαμορφώσουμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Πάντως εδώ είναι όλοι. Τώρα είναι όλοι εδώ. Μάλιστα, ένα λεπτό δώστε μου, λέει η κυρία Βέμπερ. Θέλω να εξηγήσω ότι έπρεπε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη λόγω του ατυχήματος της κυρίας Μάκιντάιρ που έσπασε το πόδι της και που μας ανάγκασε να αλλάξουμε όλη την ημερήσια διάταξη. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη και την ψηφοφορία στις 11. Ξέρετε πως είναι αυτά, όποτε έχουμε ψηφοφορία μας δεσμεύει. Εγώ θέλω να εκφράσω ευχές για την κυρία Μακιντάρ για περαστικά στην ψηφοφορία ξέρουμε ότι θα έρθουν όλοι. Και το να πιέζομαι να περάσουμε στην ψηφοφορία επειδή κάποιος έχει να κάνει κάτι άλλο μετά ή θέλει να προλάβει την πτήση του, αυτές οι πιέσεις ε, είναι μεγάλες και τρέχουμε προσπαθώντας να ανταποκριθούμε. Τώρα ε, ο κύριος Σόιερ, από το, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου για τα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Μέσων, ήρθε Αφού λοιπόν ο εκπρόσωπος του, Ευρωπαϊκού, του ε, Ινστιτούτου είναι εδώ και έχουμε και την κυρία Βέμπερ εδώ και έχουμε και τους σκιώδεις εισηγητές εδώ, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης ε, για τις πρότυπες διευθετήσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σόιερ που είναι ο εκπρόσωπος, όπως είπαμε, του Ινστιτούτου του Ευρωπαϊκού Δικαίου για τα Μέσα Ενημέρωσης. Θα παρουσιάσει ο κύριος Σόιερ τα ευρήματα μιας μελέτης που ζητήθηκε από τη ΛΥΜΠΕ με τίτλο «Το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση δίκαιο και πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της και μετά θα μιλήσει η κυρία Βέμπερ και θα εξετάσουν τα μέλη την έκθεση. Κύριε Σόιερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στην εισηγήτρια και στους ε, ευρωβουλευτές. Μου είπαν να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα που είναι τα γερμανικά και επιθυμώ να περάσω στα γερμανικά τώρα. Σήμερα το πρωί θα σας ε, κάνω μια σύντομη παρουσίαση για τα βασικά πορίσματα της μελέτης ε, που μας εξουσιοδοτήσατε να κάνουμε για την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στα κράτη-μέλη και το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Ε, έχετε το, τα περιεχόμενα μπροστά σας. Ε, αρχίζω παραπέμποντας σύντομα, αναφέροντας σύντομα τις τρεις διαφορετικές εκδοχές που υπάρχουν στη μελέτη. Έχουμε την πλήρη παρουσίαση με 710 σελίδες και από αυτή αυτό το, την πλήρη έκθεση ε, συναγάγαμε μία σύνοψη με τα σημαντικότερα πορίσματα και κατά δεύτερον μία άλλη σύνοψη που παρουσιάζει τις εκθέσεις των χωρών που συντάχθηκαν από τους ε, ε, ε, εθνικούς εκπροσώπους, τους ειδικού. Σήμερα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα περιοριστώ στα σημαντικότερα πορίσματα και αν έχετε ενδιαφέρον για να δείτε τα αποτελέσματα της κάθε χώρας ή κάποιας χώρας, μπορείτε να δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες, να ψάξετε να βρείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες για κάποια χώρα. Τώρα, για τη μεθοδολογία μας, για τη μελέτη, καταρχήν μελετήσαμε τις ε, σημαντικότερες ε, καινούριες εξελίξεις στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τότε που το 2004 είχε γίνει η πρώτη μελέτη για το ζήτημα αυτό, πάλι για το Κοινοβούλιο. Κατόπιν τούτου επεξεργαστήκαμε ένα ερωτηματολόγιο για το οποίο στείλαμε στους εθνικούς εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη και που αυτό αποτέλεσε τη βάση για την κατάρτιση των εθνικών εκθέσεων. Τα σχέδια των εθνικών εκθέσεων τα συζητήσαμε εντατικά με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες και όπου χρειαζόταν ζητήσαμε διευκρινήσεις, ε, συμπληρωματικά στοιχεία ιδιαίτερα εκεί όπου δίσταζαν οι εθνικοί ε, αντιπρόσωποι να εκφράσουν συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης στις χώρες μέλη. Αφού τέλειωσε και αυτό το στάδιο, προχωρήσαμε να κάνουμε μια συγκριτική ανασκόπηση, μια συγκριτική ανάλυση, η οποία ε, ολοκληρώθηκε με ένα ε, άλλο σημαντικό κομμάτι της μελέτης που είναι τα ευρωπαϊκά benchmarks, τα ε, συγκριτικά σημεία αξιολόγησης. Εκεί βλέπετε τα σημαντικότερα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία των ΜΜΕ και των πολιτών και είναι ο πύχης αν θέλετε, το μέτρο μέτρησης και είναι και ε, μια επιταγή για τη λειτουργία των ΜΜΕ στα κράτη-μέλη. Και με βάση αυτό συναγάγαμε σειρά συστάσεων για τις περαιτέρω διαδικασίες και εξελίξεις. Σύντομα για την κατάσταση στα κράτη-μέλη, σε επίπεδο συνταγματικό, σε όλα τα κράτη-μέλη, υπάρχει η ελευθερία έκφρασης της γνώμης και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και η ελευθερία της αναζήτησης πληροφοριών και της απόκτησης πληροφοριών. Αυτό όμως δεν ισχύει με τον ίδιο ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, πώς μπαίνει στην αγορά κάποιος πάροχος υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι έκπληξη να σας πω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ε, διαχωρισμός μεταξύ της πρόσβασης στις ραδιοφωνικές εκπομπές και στον τύπο. Ε, με αφορμή την πρόσβαση στην αγορά γίνεται μια εξέταση στα κράτη-μέλη για να δούμε ε, σε ποιο βαθμό υπάρχει συγκέντρωση ιδιοκτησίας των ΜΜΕ αλλά η έρευνα αυτή δεν γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί όπου προβλέπεται αυτό από τον νόμο και υπάρχουν οι σχετικές ρυθμίσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τη διαφάνεια των ιδιοκτησιακών σχέσεων και τη... τον αριθμό ιδιοκτησίας ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τα δημόσια μέσα, ε, αυτά που είναι μια δημοσίου δικαίου, θα πρέπει να ε, είδαμε πώς μπορούν να ε, διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, εάν έχουν επαρκή χρηματοδότηση, αν η χρηματοδότηση αυτή είναι ενδεδειγμένη για να στηρίξει την ανεξαρτησία τους, τα καθήκοντα των δημοσίων μέσων πώς περιγράφονται και αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι για το πώς ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους αυτοί, χωρίς να επισέλθουμε βέβαια στην ελευθερία, χωρίς να επισέρχονται στην ελευθερία των ΜΜΕ. Εδώ σε κάποια κράτη-μέλη εξακολουθούν να υφίστανται ελλείμματα. Επίσης από μια σειρά από κράτη-μέλη ενημερωθήκαμε ότι το νομικό πλαίσιο για τους εποπτικούς φορείς των ΜΜΕ είναι ανεπαρκής και πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα και σε σχέση με την ανεξαρτησία των παρόχων αλλά και την ανεξαρτησία από τους πολιτικούς και την πολιτική γενικότερα. Η καθ' αυτό, η κατεξοχήν δραστηριότητα των ΜΜΕ αυτονοήτως εξαρτάται κυρίως από το πώς θα καταφέρουμε το ρόλο των ΜΜΕ να τον διασφαλίσουμε τον ρόλο τους ως watchdog. Και εδώ από τις εκθέσεις των κρατών μελών προκύπτει μια σειρά ελλημάτων που δεν ε, προσδιορίζεται και δεν οφείλεται στην ομοθεσία την υφιστάμενη, αλλά έχει περισσότερο να κάνει με την πρακτική εφαρμογή των νόμων για την ελευθερία των ΜΜΕ. Είναι αδιαφανές σε πολλές περιπτώσεις σε ποιο βαθμό υπάρχει προστασία των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά την επιγραμμική δραστηριότητα των δημοσιογράφων online και γενικά το επαγγελματικό καθεστώς του δημοσιογράφου δεν ορίζεται παρά μόνο σπάνια, άρα και από εκεί προκύπτουν κάποιες ασάφειες και αβεβαιότητες. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης σπάνια χρησιμοποιούν το μέσον ε, που προβλέπει θετικές προδιαγραφές που θα εκδίδονται για τα ΜΜΕ, για τις μειονότητες, για τον πολιτισμό που όπως προβάλλονται αυτά στα ΜΜΕ. Εκτός από το σύστημα του, των δημοσίων ραδιοφωνικών σταθμών, σπάνια υπάρχουν συστήματα τα οποία εξυπηρετούν στη χρηματοδότηση περιεχομένων ε, που συνδέονται με κάποια ε, γενικότερη αξία, μια κοινή, ένα κοινό αγαθό. Ε, στο ΜΜΕ, στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στον τομέα του τύπου ε, υπάρχουν κάποιες τέτοιες δραστηριότητες, αλλά σε πολλές χώρες οι κώδικες που υπάρχουν δεν εφαρμόζονται όπως πρέπει και αυτό σημαίνει ότι πολλοί ε, δεν, πολλοί ε, πάροχοι ε, δεν σέβονται τις προδιαγραφές. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσα από τα ΜΜΕ μόνο εάν αυτά μπορούν να είναι ευρέως διαδεδομένα. Ζητήσαμε να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν εμπόδια για τη διάδοση των ΜΜΕ ή αν υπάρχουν και από την άλλη πλευρά δυνατότητες διευκόλυνσης της διάδοσης ηλεκτρονικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος. Ξέρουμε ότι παρά το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην προσέγγιση ραδιοφωνικών συχνοτήτων στο ραδιόφωνο, πρόσβαση σε πλατφόρμες στο ραδιόφωνο και ξέρουμε ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν δυσκολίες και για τα προϊόντα του τύπου που δεν βρίσκουν εύκολα τα, το δρόμο για τα σημεία διανομής και τα περίπτερα. Έτσι θα έπρεπε να δούμε και να ελέγξουμε το δίκαιο ανταγωνισμού που μπορεί να γίνει όμως ε, μπορεί μόνο όμως να γίνει και να αποτρέψει δυσκολίες εκ των υστέρων, όχι να τις προβλέψει και να τις αποτρέψει εκ των προτέρων. Τώρα, το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία, ιδιαίτερα πρόσβαση στην πληροφορία που προέρχεται από κρατικές δημόσιες πηγές. Εδώ συχνά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλήρης νομοθεσία για το θέμα αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη μπήκαν τώρα σε αυτή τη διαδικασία θέσπισης και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης σημαντικό ήταν να δούμε αν ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί από ποιον προέρχεται η πληροφορία που παίρνει στα ΜΜΕ. Δηλαδή, εδώ είναι ένα θέμα διαφάνειας των ε, σχέσεων ιδιοκτησίας και του πραγματικού ε, ιδιοκτήτη των μέσων. Εδώ πράγματι υπάρχει μια σειρά από ελλείμματα. Για τα, τους δημόσιους ε, φορείς, ΜΜΕ, έχει ενδιαφέρον να ξέρει ο πολίτης ε, τι ε, επιδόσεις έχει μέσα στην κοινωνία, οπότε θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στους δημόσιους φορείς και ποιος προσπαθεί να δημοσιεύει τέτοιου είδους εκθέσεις. Και εδώ υπάρχει διαφορετική κατάσταση στα 27 κράτη-μέλη. Κατά κανόνα δεν υπάρχουν δυσκολίες για τους πολίτες να βρουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των ΜΜΕ εκτός αν είναι οικονομικές οι δυσκολίες και γι' αυτό μια σειρά από κράτη-μέλη ε, προσφέρουν συστήματα βοηθητικά ούτως ώστε οι εισοδηματικά ε, αδύναμοι πολίτες παρόλα αυτά να έχουν πρόσβαση στα ΜΜΕ. Το τελευταίο θέμα που μας απασχόλησε αφορά το πώς, με ποιο τρόπο μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στην διαμόρφωση και τη δημιουργία των περιεχομένων των ΜΜΕ. Έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να ε, επικρίνουν τις εκπομπές ή μπορούν εκ των προτέρων να επηρεάζουν τα περιεχόμενα εκφράζοντας επιθυμίες, αιτήματα κλπ. Και εκεί πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ελάχιστα συστήματα ε, όπου οι πολίτες μπορούν είτε άμεσα είτε με εκπροσώπους των συμφερόντων τους να παρεμβαίνουν στα ΜΜΕ. Τέλος, η κατάσταση της αγοράς μιμιέ δεν θα σας εκπλήξει αν σας πω ότι δεν θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω λεπτομερείς παρατηρήσεις. Περιορίζομαι να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και αυτό δεν έχει πάντοτε να κάνει με την οικονομική κατάσταση στην κάθε χώρα. Μπορεί να είναι η εξήγηση και πολιτιστική, πολιτισμική. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αγορά, είτε στον τύπο, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, κατά κανόνα δεν επιτρέπει να ε, συμπεράνομαι αν έχουμε πλουραλιστικό περιεχόμενο ή ποικίλο περιεχόμενο και αν ο πολίτης έχει περισσότερες προσφορές ή αν θα ήταν, είναι καλύτερα ή αν έχει λιγότερους ε, ε, παρόχους που όμως είναι πιο οικονομικά ισχυροί. Ε, ένα άλλο θέμα είναι η, θέση των δημοσίων ΜΜΕ και ο ρόλος που πρέπει να παίξουν για να αντισταθμίσουν την παρουσία των εμπορικών παρόχων. Το έργο τους καθίσταται ε, δυσκολότερο διότι αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις αλλά πολλές φορές υποφέρουν και λόγω των πιέσεων από τους πολιτικούς. Το ενδιαφέρον των εθνικών αντιπροσώπων εστιάζεται στη βελτίωση της ε, νομικής κατάστασης ε, και της εφαρμογής του νόμου αλλά και της παρεμβάσεις ε, που περιμένουν να γίνουν, ε, για παράδειγμα, για την ε, πολιτιστική ποικιλομορφία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή του εθνικού δικαίου για τα ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της απόφασης του ε, Στρασβούργου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το άρθρο 10 ειδικότερα. Σε πολλές εθνικές εκθέσεις αναφέρεται το θέμα της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, την αυξανόμενη συγκέντρωση και την έλλειψη διαφάνεια σχετικά με τους πραγματικούς ε, ιδιοκτήτες. Ε, τώρα, τα σημαντικότερα πορίσματα σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη σημασία του για τα ΜΜΕ και την ε, ελευθερία πληροφόρησης. Ε, στο άρθρο 11 του Θεμελιώδους Χάρτη και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αυτά είναι τα σημαντικά, οι βασικές ελευθερίες, το δίκαιο ανταγωνισμού, αλλά και η πολιτισμική ρήτρα της ε, ε, αναφοράς για τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης. Επίσης, το παράγωγο δίκαιο, ιδιαίτερα η οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, το δίκαιο τηλεπικοινωνιών, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά και οι ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι σημαντικές εδώ, και τέλος, πολύ σημαντικό, η νομολογία των, του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο, των δικαστηρίων στο Λουξεμβούργο. Σημαντικό, ε, το σημαντικό συμπέρασμα παραμένει αμετάβλητο ότι το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, είναι ο βασικός πυλώνας ε, για την ελευθερία των ΜΜΕ στην Ευρώπη και για την ελευθερία πληροφόρησης δεν εκπλήσει σε αυτά τα πλαίσια η απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και χαιρόμεθα διότι το άρθρο 11 του, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προβλέπει ότι ε, σημειώνονται, ε, ε, πρέπει να σημειωθούν εξελίξεις. Αναφέρεται ρητά από το Δικαστηρίο ότι τα κράτη τα οποία είναι οι θεματοφύλακες της ποικιλομορφία σε, τελευταία ανάλυση τα κράτη ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν όλα τις ίδιες υποχρεώσεις εδώ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το δημόσιο, τα δημόσια μήμια, το δημόσιο ραδιόφωνο, το οποίο πρέπει να την χάνει επαρκούς χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ε, περιλαμβάνουν και έχουν μέτρα τα οποία θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να λαμβάνονται υπόψη, να λαμβάνονται περισσότερα υπόψη. Επίσης, ε, το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό έχει να κάνει με τις αρχές της εξουσιοδότησης και της επικουρικότητας Επίσης, ε, ε, ε, μηχανισμοί εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά θα πρέπει να έχουν τέτοιο προσανατολισμό ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Όμως φαίνεται ότι ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακόμα επαρκώς σαφές με ποια μορφή η αρχή του κράτους δικαίου και η αρχή της δημοκρατίας ως υποχρεωτικές αξίες για όλα τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να επηρεάσουν την διαμόρφωση ε, της λειτουργίας των ΜΜΕ και τις τάξεις που επικρατεί σε αυτά. Ακόμη δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη απάντηση εκτός από το άρθρο 11 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δούμε εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες από την εφαρμογή του άρθρου. Έχουμε την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου είναι εκείνο το οποίο ε, ε, ενσωματώνει το άρθρο 11 ε, του χάρτη και φροντίζει και επιμένει για την σωστή εφαρμογή του. Τέλος, εις ό,τι αφορά τις συστάσεις που μπορούμε να κάνουμε με βάση τα ευρήματα αυτά, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι θεωρούμε σημαντικό να βρεθεί ένα μόντους βιβέντη ε, με το Συμβούλιο της Ευρώπης γιατί αυτό θα αποφέρει ωφέλη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ορίσουμε περισσότερο την συμπληρωματικότητα των δύο οργανισμών στον τομέα της ελευθερίας του δικαίου ε, για τα ΜΜΕ και της ελευθερίας έκφρασης. Παρόμοια ε, σύσταση ισχύει και για άλλα διεθνή φόρα με τα οποία ε, μπορεί να δραστηριοποιηθεί από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε θέματα της πολιτικής των συχνοτήτων, στο το διαδίκτυο κλπ. Πάντοτε συνεργαζόμενοι με τα αντίστοιχα ε, Φαίνεται ότι Χρειάζεται υψηλότερος βαθμός συνοχής μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν τα ΜΜΕ και που είναι καθοριστικές για το δικαίωμα των πολιτών να ε, ζητούν πληροφορίες και ενημέρωση. Με όλες, σε όλες τις δραστηριότητες των ΜΜΕ είναι σημαντικό πιστεύουμε να ακολουθηθεί η προσέγγιση του Κοινοβουλίου, δηλαδή ε, να ε, δούμε τα μέσα ως προϊόντα ζωτικής δημοκρατικής σημασίας και που έχουν πολιτισμική αξία και αποτελούν και παράγοντα ε, σημαντικό για τις οικονομίες. Αυτός ο διτός χαρακτήρας δεν αποτελεί αντίθεση, αντίθετα μπορεί να ε, οδηγήσει σε αμοιβαία γονιμοποίηση. Τώρα γίνεται ενημέρωση ε, των πληροφοριών μέσα από τη μελέτη αυτή. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό για την ελευθερία του ΜΜΕ να υπάρχει ε, μια σταθερότερη βάση και εδώ να φροντίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στο μέλλον. Πρέπει να διασφαλιστεί ε, ότι οι πληροφορίες ε, θα προέρχονται πάντα από μια αξιόπιστη ε, στιβαρή βάση. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα επίπεδο όπου πολλοί οργανισμοί, ιδρύματα, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται πια με τα θέματα αυτά. όμως εκείνο που λείπει είναι ότι δεν υπάρχει συνεργασία επαρκής των διαφόρων φορέων, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνει για παράδειγμα ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Βιέννη, για να πω έναν, ε, και πώς μπορούμε έτσι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικότερο τρόπο τους λίγους σπόρους που διαθέτουμε. Τέλος, ε, θα πρέπει να δούμε αν η μέχρι τώρα ε, δομή του σχετικού άρθρου στην Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σωστά διατυπωμένο. Δηλαδή, ε, κάθε εναρμόνιση και κάθε δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα έπρεπε να ε, αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα ή υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθούν εδώ κάποιες προσεγγίσεις. Τέλος, συστάσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη πολιτική ε, των ε, ΜΜΕ. Θα έπρεπε πιστεύουμε να σκεφτούμε αν χρειάζεται, αν είναι ενδεδειγμένο να ζητήσουμε επίσημα από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ε, οδηγίας ή κάποιο άλλο μέσο σχετικά με την ιδιοκτησία και την συγκέντρωση των ΜΜΕ και να ε, θεσπίσει τουλάχιστον κανόνες διαφάνειας που θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, εδώ ε, συζητούμε μία επέκταση του πεδίου εφαρμογής και αν είναι δυνατόν με αυτό το μέσον το οποίο προβλέπει ε, δικαίωμα ε, κατά αντιπαράσταση ε, ή αναφέρεται σε δικαιώματα των πολιτών για ενημέρωση σε σημαντικά γεγονότα, να δοθούν περισσότερες διασφαλίσεις για την ελευθερία των μέσων και την ελευθερία και το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση. Τώρα, στο παράγωγο δίκαιο πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό λαμβάνοντα υπόψη την εξέλιξη των ηλεκτρονικών μέσων και της τηλεόρασης και της εξέλιξης του διαδικτύου, να ξαναδούμε την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να δούμε ιδιαίτερα τον ρόλο των διαμεσολαβητών, των ενδιαμέσων και επίσης να δούμε και την ε, ε, νομοθεσία που διέπει τα προϊόντα για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν κάποια ε, θέματα που θα έπρεπε να ε, βελτιώσουμε σε ό,τι αφορά την ελευθερία των ΜΜΕ και τα δικαιώματα των πολιτιωτών. Η Apple, ας πούμε, αποφασίζει τι καρτούν θα προβληθεί σε ένα iPhone στην ε, Ευρώπη ή σε ένα κράτος μέλος. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την ελευθερία ε, των ΜΜΕ και τα δικαιώματα των πολιτών. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε σκεφτεί όταν μιλούσαμε για την τυποποίηση και άλλα θέματα παρόμοια. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενδιαφερθεί ε, στη, για τη συζήτηση σχετικά με την ε, ουδετερότητα και την παραγωγή ε, των περιεχομένων των ΜΜΕ και θα πρέπει να δούμε πώς ε, παράγεται και διαδίδεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων των ΜΜΕ. Επίσης σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον για τη μελλοντική ε, πολιτική των συχνοτήτων. Τέλος, αυτό το λένε και οι εκθέσεις των κρατών μελών, φαίνεται ότι το copyright και τα προστατευόμενα δικαιώματα σε ε, νοσιακό επίπεδο θα πρέπει να αναθεωρηθούν και μάλιστα αρκετά σύντομα. Βέβαια αυτό είναι ένα δύσκολο αίτημα εις ό,τι αφορά τον περιορισμένο χρόνο της θητείας που έχει απομείνει. Ε, ε, έφτασα στο τέλος της παρουσίασής μου και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Βεβαίως είναι δύσκολος ο στόχος. Κανείς δεν έχει πει ότι είναι εύκολος. Βρισκόμαστε στο μέσο της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα βεβαίως θα δώσω το λόγο στην κυρία Βέμπερ ε, έτσι ώστε να παρουσιάσει την έκθεση και μετά ε, καταγράφουμε αυτούς που θέλουν να πάρουν το λόγο μετά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόγερε για την παρουσίασή του αλλά και για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε έτσι ώστε να είναι σήμερα μαζί μας. Πιστεύω ότι δύσκολα θα βρει κανείς πιο κατάλληλο χρόνο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έκθεσης και την παρουσίαση των συστάσεων τη στιγμή που έχουμε να ετοιμάσουμε αυτήν την έκθεση. Πολλές από τις συστάσεις σας οπωσδήποτε μέσω των τροπολογιών θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην έκθεση αυτή. Όπως γνωρίζετε όλοι, πρόκειται για ε, ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Γι' αυτό δεν θα με εκπλήξει αν ο αριθμός των τροπολογιών είναι εντυπωσιακά μεγάλος. Την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, Πολλά ψηφίσματα και συστάσεις έχουν εκπονηθεί και ε, εγκριθεί από τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΣΑ, ε, ακόμα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι μία δόκιμη ερώτηση είναι γιατί χρειαζόμαστε κι άλλη έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας με το ίδιο θέμα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με δύο άλλα ερωτήματα. Είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση των ΜΜΕ στα κράτη-μέλη. Μας αρέσει το, το, το, το τοπίο που βλέπουμε στα κράτη-μέλη. Και η άλλη ερώτηση. Είμαστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις που μας έχει δώσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποτεδήποτε υπήρχαν σημαντικά σημάδια ε, ε, μη ελευθερίας των ΜΜΕ σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μάλλον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, να διασφαλίσουμε ότι η ελευθερία των μέσων και ο πλουραλισμός γίνονται απολύτως σεβαστά, όπως ακριβώς ρητά αναφέρεται στο άρθρο 11 ε, της ε, Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας έφτασε η ώρα να συζητήσουμε και τις εξουσίες οι οποίες απορρέουν από το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ε, συνθήκης θεμελιωδών δικαιω... της, ε, της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μερικά πράγματα μόνο θα αναφέρω, δεν θα αναλύσω σε βάθος την κατάσταση. Ευελπιστώ ότι μέχρι το τέλος ε, ε, μέχρι την ολοκλήρωση δηλαδή της ε, συζήτησης και την ψήφιση της έκθεσης ότι θα έχουμε στο τέλος έναν κατάλογο ε, με αυτά που πρέπει να κάνουν οι χώρες μέλη και έναν άλλο κατάλογο με αυτά που δεν πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και ότι θα υπάρχουν και αυτοί οι ίδιοι κατάλογοι, οι ίδιες λίστες και για την Κομισιόν. To do και not to do. Έχουμε και μια οικονομική κρίση, μην το λησμονούμε, η οποία έχει πάρα πολύ κακές επιπτώσεις στα μέσα ενημέρωσης και στην ε, επιβίωση των μέσων ενημέρωσης και στην ελευθερία των μέσων και ε, στην ελευθερία των δημοσιογράφων κλπ αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες νομοθετικά δεσμευτικοί ε, έτσι ώστε να μην υφίστανται χειραγώγηση τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι. Για... Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσουν να επιτύχουν το αποτέλεσμα αυτά τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν ο κατάλογος με αυτά που δεν πρέπει να γίνονται, η not to do list, θα πρέπει να περιέχει πολλά πράγματα. Ας πούμε, να μην χρησιμοποιείται άσχημα η νομοθεσία ε, της κρατικής ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας. να μην χρησιμοποιείται η κρατική προπαγάνδα για να στηρίζονται αυτά τα μέσα ενημέρωσης, αυτές οι κυβερνήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους. Υπήρξαν φήμες ε, πολύ καιρό, αλλά τώρα πλέον είμαστε σίγουροι ότι στον κατάλογο το not to do θα πρέπει να αναφέρεται ότι ε, βάση νομοθεσίας ε, θα πρέπει να απαγορεύεται ε, σε μυστικές υπηρεσίες ε, να παριστάνουν τους δημοσιογράφους και να προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες κάνοντας ότι είναι δημοσιογράφοι. Είχαμε φήμες πολύ καιρό, αλλά τώρα σε μερικές περιπτώσεις έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία. και βεβαίω τον κατάλογο των ε, σωστών πρακτικών που βεβαίω δεν θα έχουν τη μορφή καταλόγων στην έκθεση ε, θα πρέπει να πούμε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν με κάθε τρόπο και με κάθε νομική στήριξη ε, την ελευθερία, την ανεξαρτησία των ε, ε, μέσων ενημέρωσης ε, και εκεί το θέμα της ιδιοκτησίας των μέσων είναι πολύ σημαντικό. Το, τους τελευταίους μήνες είχα πολλές συναντήσεις και πρέπει να σας πω ότι όλες οι ενώσεις, οι ομοσπονδίες δημοσιογράφων, είτε πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες, για ιδιωτικό τομέα, για ιδιοσιογραφικά πρακτορία κτλ όλοι θέλουν ε, ε, διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο και ότι τα προσκόμματα είναι πολλά. Ναι, αλλά αν ξεκινήσουμε σηκώνοντα τα χέρια λέγοντα Α, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, αυτό είναι ανεπίτευκτο στόχο, τότε δεν έχει έννοια να ασχολούμαστε με αυτό. Τότε γιατί προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την το οργανωμένο έγκλημα ή την ε, ε, λογοκρισία ή, οποιασδή, ή οτιδήποτε άλλο ή τη διαφθορά. Να μην είμαστε υποκριτικοί και να λέμε ότι μόνο στο θέμα τη δημοσιογραφία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα νέο νομικό περιβάλλον ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων βεβαίως είναι νομικός δεσμευτική. Αλλάζει το τοπίο ήδη. Αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλά κουράστηκα πια να λέω και να επαναλαμβάνω εδώ στο Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να ε, τίθεται σε εφαρμογή σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της Συνθήκης Λειτουργίας ε, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι ε, η συνθήκη υπάρχει και ότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι παράγωγο δίκαιο. Αυτό το έχει πει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό και προσδοκώ να το δω να γίνεται πραγματικότητα είναι ε, η ε, εποπτεία, το monitoring και η αιτήσια αναφορά. Και εδώ μιλάμε για σεβασμό των αρχών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα όργανο κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά θα μπορούσε να είναι και το Κέντρο για τον Πλουραλισμό και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης. Γνωρίζω ότι υπάρχουν νομικές δυσκολίες, ας το πούμε έτσι. Πάντως να υπάρχει ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα πρέπει να αναφέρεται, να κάνει αναφορές για τα θέματα αυτά κάθε χρόνο σε αιτήσια βάση με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένα ονόματα. Όχι γενικά και αόριστα. Ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει προβλήματα με τα μέσα ενημέρωση σε κάποιες χώρες μέλη. Πριν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 7, θα πρέπει καλύτερα να προβλέπουμε να δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών, με συγκεκριμένα παραδείγματα κακών πρακτικών, λαθών κτλ. Έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μέσα πίεσης ε, να έχει την δυνατότητα να δείξει αυστηρότητα απέναντι στην ε, χώρα γιατί μέχρι τώρα είναι ε, σιωπηρή και υπερβολικά ντροπαλή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσέγγιση που έχει απέναντι στα κράτη-μέλη αυτά που παραβατούν. θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, ένα ευρωπαϊκό σώμα για την ε, ρύθμιση ε, του κλάδου. Αυτό είναι εύκολο γιατί απορρέει εύκολα από την οδηγία και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το επιτύχουμε. Πολύ γρήγορα. Θέλουμε, χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν χρειαζόμαστε. Έστω και αν σε ορισμένα προηγούμενα ψηφίσματα ε, στο Κοινοβούλιο γινόταν μια τέτοιου είδους αναφορά. Όμως, ε, συνάντησα πάρα πολλές οργανώσεις ε, δημοσιογράφων, πάρα πολλές ομοσπονδίες κτλ. Όλοι λένε δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω νομοθεσία γι' αυτό. Όχι γιατί υπάρχει αρχή της επικουρικότητας μόνο, αλλά και γιατί η πραγματικότητα στην κάθε χώρα διαφέρει από, από χώρα σε χώρα, συγγνώμη, διαφέρει υπάρχουν και κάποιες πολιτιστικές ε, παραδόσεις ε, που θα ήταν κρίμα ε, να σταματήσουν λόγω της κεντρικής αυτής νομοθεσίας. Μιλήσουμε όμως ότι υπάρχει και πρωτοβουλία πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων από το τομέα των μέσων για άμεση εμπλοκή των πολιτών σε αυτά. Στην ακρόαση της 6ης ε, Νοεμβρίου θα συζητηθεί και το θέμα αυτό. Και μετά την ακρόαση ακριβώς ε, έχουμε προβλέψει και κάποιες μέρες ακόμα πριν ε, την λήξη της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών γιατί θα αντλήσουμε και από εκεί πολύτιμες πληροφορίες. Έχουμε επίσης την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΧΑΛΤ. <clears throat> Και θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούμε όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία στην διάθεσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον νοτάριο της Άλντε για όλη την πολύτιμη βοήθεια που μου έδωσε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέμπερ, λέει ο Πρόεδρος. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση, από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος Μπουζούτιλ. Ευχαριστώ. Παρεμβαίνω εξ του Σκιώδους, του κυρίου Μαρινέσκου σκιώδους εισηγητού του ΕΛΚ που έπρεπε να επιστρέψει στην εκλογική του περιφέρεια σήμερα. Ευχαριστώ καταρχήν την κυρία Βέμπερ για το σχέδιο έκθεσης που λέει σαφώς και, και πρέπει να πω ότι το ΕΛΚ θεωρεί την έκθεση πολύ καλή βάση και πολύ ισορροπημένη έκθεση και την εκτιμούμε όπως της αξίζει. Υπάρχουν δύο βασικά θέματα που θέλω να θέσω. Το πρώτο αναφέρθηκε ιδιαίτερα από την ίδια την κυρία Βέμπερ πριν από λίγο και αφορά τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε αυτά τα θέματα, σε ποιο βαθμό μπορούμε να εφαρμόζουμε το χάρτη της Ένωσης εδώ, σε ποιο βαθμό μπορούμε να ζητούμε από την Κομισιόν να νομοθετεί και αν είναι εδώ εκπρόσωπος της Κομισιόν, ίσως θα έπρεπε να παρέμβει στη συζήτηση αυτή και να μας πει τι ποια θεωρεί ότι είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλετε σε αυτό το τομέα. Εγώ νομίζω ότι ο χάρτης της Ένωσης δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε αυτόν τον ε, τομέα γιατί ο χάρτης της Ένωσης δεν αφορά ειδικά το, τα τεκτενόμενα στα κράτη-μέλη, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στα κράτη-μέλη ρυθμίζονται από άλλε συμβάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ χάρτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τα θεσμικά όργανα και το ενωσιακό δίκαιο και την εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει αναφορά στην πρόταση νομοθετική πρωτοβουλία στο σημείο, στην αιτιολογική σκέψη F. Δεν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα, αλλά και πάλι πρέπει η Κομισιόν παρακαλώ να μα πει αν γίνεται η Κομισιόν, γιατί είναι άσκοπο να επαναλάβουμε τα ίδια κάθε λίγο και λιγάκι χωρίς να ξέρουμε ακριβώς εάν υπάρχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο. Αν έχουμε την αρμοδιότητα, μάλιστα να πιέσουμε την Κομισιόν να, υποβα... να αναλάβει πρωτοβουλία. Αν δεν γίνεται όμως πρέπει να το πούμε άπαξ και διαπαντός και να τελειώνουμε. Το ίδιο ισχύει σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων στα κράτη-μέλη και τι γίνεται τότε. Βεβαίως αυτά πρέπει να είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν, αλλά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, για να ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε πρέπει να ξέρουμε ποιος μηχανισμός θα εφαρμοστεί. Είναι άσκοπο να ζητάς από κάποιον να να, να του ζητάς να αντιμετωπίσει την παραβίαση αν αυτός ο κάποιος δεν μπορεί, δεν έχει την αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο. Να ξέρουμε λοιπόν ποιος μηχανισμός ισχύει, πρέπει να ισχύει και να εφαρμόζεται σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου παραβίασης της ελευθερίας των μημιών. Παρομοίως, στην παράγραφο 10 υπάρχει έκκληση για την δημιουργία Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Φορέα για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που θα πρέπει να έχει και εξουσίες επιβολής κυρώσεων. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνθήκες δηλαδή δίνουν την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει μια τέτοια ομάδα. Εγώ θα ήθελα να απαντηθεί αυτή η ερώτησή μου πριν, ε, ε, πριν αποφανθώ οριστικά. Τέλος, ένα σημαντικό θέμα που, πια, που είναι η ψυχή και η καρδιά της ελευθερίας των μέσων, δηλαδή η ποιότητα της δημοσιογραφίας και των δεοντολογικών προτύπων στη δημοσιογραφία που πρέπει να περιλαμβάνει την αξία της ακαιρεότητας επαγγελματισμού, ανεξαρτησίας και προφανώς και την εφαρμογή κωδίκων συμπεριφοράς. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι στα πλαίσια της δικής μας αρμοδιότητας και εντολής να νομοθετούμε εδώ, αλλά σε μια έκθεση πρωτοβουλίας θα ήταν ίσως καλό να συμπεριλάβουμε και μία παράγραφο που θα αναφέρεται στην σημασία της ακαιρεότητας και της δεοντολογίας στη δημοσιογραφία ως πυλώνα ανεξαρτησίας και πλουραλισμού στα ΜΜΕ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κόντς, ευχαριστώ πολύ. Ε, σκιώδης από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τον κύριο Σόιερ επίσης για την παρουσίασή του και την ε, εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Θυμάμαι πώς άρχισε η δουλειά αυτή. Κάποια στιγμή η Επιτροπή Λίμπε είχε την εντύπωση ότι θα έπρεπε να θέσουμε ελάχιστε προϋποθέσεις για την ελευθερία και τον πλουραλισμό των ΜΜΕ. Και πολλά έγιναν από τότε. Εμείς συνεχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο θέμα αυτό. Γνωρίζουμε όμως ότι η Νέλη Κρούσα που είναι υπεύθυνη, από την υπεύθυνη επίτροπος για τα οπτικοακουστικά σύστησε ένα φορέα που επίσης, που δουλεύει επίσης πάνω σε αυτά τα θέματα, χωρίς συστάσεις. Και πριν από λίγες μέρες η Κομισιόν δέχτηκε μια πρωτοβουλία πολιτών για τον πλουραλισμό των ΜΜΕ, που είναι άμεση απάντηση στο θέμα ή στο δίλημα που υπάρχει πάντα όταν συζητάμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν και αν γίνει δεκτή η πρωτοβουλία των πολιτών, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει το θέμα. Είπατε επίσης ότι είναι πολύ κατακαιρματισμένο το ενωσιακό πλαίσιο. Από τη μία πλευρά συστήνει έντονα η έκθεση των συντονισμό και την εναρμόνιση σε κάποιους τομείς, σοβαρή παρακολούθηση, ε, συμφωνούμε εδώ απόλυτα. Αλλά σε αντίθεση με τον κύριο Μπουσουτή εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ε, καταθέσουμε ένα κατάλογο ελάχιστων προϋποθέσεων για την ελευθερία και τον πλουραλισμό των ΜΜΕ. Επίσης αναφέρατε διάφορες πτυχές των προβλημάτων. Ε, είναι ενδιαφέρον ότι τώρα έχουμε πολύ πιο πλήρη κατάλογο των προβλημάτων από ότι <laughs> κατάλογο λύσεων και συστάσεων. Αλλά είναι ευθύνη μας επίσης να δώσουμε συνέχεια στις συστάσεις. Είναι σημαντικό να ζητήσουμε από την ε, νομική υπηρεσία, όπως είπε η Ρενάτε Βέμπερ στο έγγραφο εργασίας, θα χρειαστεί να ρωτήσουμε όλες τις νομικές υπηρεσίες αλλά και την Κομισιόν πώς ερμηνεύουν τις αρμοδιότητές τους. Επίσης είναι ευθύνη μας ε, να παρουσιάσουμε και εμείς συστάσεις για ελάχιστες προϋποθέσεις και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να συνεχίσει προς την κατεύθυνση μιας οδηγίας. Δεν μπορεί να έχουμε κανονισμό, στιβαρό και λεπτομερή, αλλά ε, ένα πλαίσιο για την ελευθερία των ΜΜΕ και τις ε, ελευθερίες για τον πλουραλισμό και την ελευθερία των μέσων που θα ρυθμίζει και τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας που είναι ένα θέμα που προκύπτει ξανά και ξανά και που είναι ένα από τα δύο μεγάλα θέματα γνωρίζοντας την κατάσταση στα κράτη-μέλη Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά θαραλέοι για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα αυτά, να τους δώσουμε συνέχεια, να γίνει πρόοδος. Και βέβαια πρέπει να ελέγξουμε τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Ταυτόχρονα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι στη γνώμη μας και εγώ θα ήθελα να συνεργαστώ με τους σκιώδεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκόνς. Κυρία Ιντερβέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, αντιδρώντας αυτά που είπε ο Σάιμον Μπουσουτήλ, κάθε φορά που γίνεται κάτι που δεν θέλει μια πολιτική ομάδα, έχουμε το επιχείρημα για τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Πολλά γίνονται στην Ευρωζώνη ε, όπου είναι, υπάρχει πάρα πολύ ισχνή βάση στις συνθήκες, αν υπάρχει, και παρόλα αυτά υπάρχει πολιτική συνένεση ότι πρέπει να γίνει αυτό. Χθες μόλις η ομάδα σας υποστήριξε μια έκθεση η οποία ευτυχώς απορρίφθηκε στην Επιτροπή Γυναικών για τον περιορισμό των ΜΜΕ προκειμένου περί εικόνων γυναικών. Ε, έχουμε αρμοδιότητα να το κάνουμε αυτό. Δεν νομίζω. Γιατί λοιπόν υποστήριξε την έκθεση η ομάδα σας. Αν πιστεύουμε ότι πρόκειται για ε, ευρωπαϊκές αξίες και αν η Ένωση είναι κοινότητα αξιών, αυτός πρέπει να είναι πολιτικός στόχος. Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει νομική βάση, να φτιάξουμε βάση στη μελλοντική συνθήκη. Α μπούμε στην ουσία λοιπόν των πραγμάτων και α μην κρυβόμαστε πίσω από τι εξουσίε και τι αρμοδιότητε και ε, ψευδονομικίστικα επιχειρήματα. Θέλετε να προστατεύσετε την, ελευθερία των μέσων. Ε, να προχωρήσετε και να την προστατεύσετε. Ευχαριστώ την κυρία Ίνφελτ, ε, κυρία Ραντίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα, μετά την κυρία Γκόντ και την κυρία Ινφελτ, ε, λέει η κυρία Σαρτζεντίνη, θα ήθελα να πω και εγώ κάτι παρόμοιο. Αυτή τη βδομάδα στην ε, Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών παρουσιάστηκε μία έκθεση για, τον διερευνητικό, για τη διερευνητική ε, δημοσιογραφία σε σχέση με την απάτη με ενωσιακή χρηματοδότηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση να τη διαβάσετε. Ε, παρουσιάζει παραδείγματα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πώς η δημοσιογραφία πρόβαλε περιπτώσεις απάτης ε, με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έφερε στο φως όλα αυτά και έτσι μπορούμε να παίρνουμε περισσότερες τέτοιες πληροφορίες. Πέρα από την ελευθερία των ΜΜΕ υπάρχει και ανάγκη ευρω... τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αλλάξουν τη στάση τους προ η συζήτηση για την πρόσβαση στα έγγραφα. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα ε, θεσμικά όργανα εδώ στις Βρυξέλλες δεν θέλουν τη διαφάνεια και θέλουν να ε, παραμείνουν στην αρχή ότι όλα είναι μυστικά εκτός αν ισχύει κάτι διαφορετικό. Αντί για το αντίθετο. Μιλάμε, μιλάει για αυτούς που ε, αποκαλύπτουν ειδήσει ή την προστασία των πηγών των δημοσιογράφων και δείχνει ότι αν θέλουμε να έχουμε καλή δημοσιογραφία πρέπει να έχουμε και πολιτικούς που να είναι διατεθειμένοι να είναι διαφανείς, να προστατεύουν τη διαφάνεια και να προστατεύουν τους δημοσιογράφους. Αυτό συνδυάζεται με την τωρινή συζήτηση και την έκθεση της κυρίας Βέμπερ που συζητάμε, που είναι το αποτέλεσμα μιας σοβαρότατης συζήτησης για το, ε, για το δίκαιο των ΜΜΕ στην Ουγγαρία και αναφέρεται και σε προηγούμενες συζητήσεις ε, κατά τη θητεία αυτή, δηλαδή την κατάσταση ε, των ΜΜΕ στην Ιταλία. Το γεγονός ότι προσπαθούμε να βρούμε εργαλεία για να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τα πλουραλιστικά μέσα και την προστασία των δημοσιογράφων είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και ξανά και ξανά αρχίζουμε μια συζήτηση που λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε. Νομίζω ότι η κυρία Ίντφελτ έχει δίκιο. Πρέπει να βρούμε τρόπους, να έχουμε το δικαίωμα να παρέμβουμε. Και είμαι λίγο απογοητευμένη, διότι η Ρενάτε Βέμπερ, που το θέμα το ξέρει άριστα, Μόνο ο ακροθυγός μιλάει για το θέμα ότι το κοινοβούλιο αυτό επανειλημμένα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ψήφο κατά πλειοψηφία ότι θέλουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Το λέτε στην αιτιολογική σκέψη F, αλλά δεν το υπογραμμίζουμε μόνο, δεν το υπενθυμίζουμε μόνο, όχι. Απαιτούμε, δια, ε, ζητούμε ε, νομοθετικό, νομοθέτημα. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε για τη Ρουμανία την επόμενη φορά. Αν όμως δεν μπούμε στα κράτη μέλη, πρέπει όμως να πούμε παράλληλα στα κράτη μέλη ότι πρέπει να διορθωθούν. Αλλιώς τα παραδείγματα θα πολλαπλασιάζονται όπου θα ε, κάνουν τα μέσα να σιωπούν και ξέρουν οι πολιτικοί ότι αν ε, κάνουμε τα ΜΜΕ να σιωπήσουν, αν τα κλείσουμε τότε πάσχει η δημοκρατία. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Σόγερ για την σημερινή του παρασίαση, την οποία ε, θεωρώ πολύ χρήσιμη και για τη συστάση του. Και βεβαίω να ευχαριστήσω και την Ρενάτε Βέμπερ, γιατί πιστεύω ότι όντω η έκθεσή τη αποτελεί πολύ καλή βάση για την ε, συζήτηση. Βεβαίω ε, θα υπάρξουν πολλέ τροπολογίε. Θα βάλω και εγώ τα δυνατά μου έτσι ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Συμφωνώ με την Σόφι Βεβαίως η αντιπροσωπεία μου πάντα ε, είναι πάρα πολύ προσεκτική όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας και ενδεχόμενη παραβίασή της. Αλλά νομίζω ότι στην προκείμενη περίπτωση Νομίζω, λέω, ότι υπάρχουν πολλές ε, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ανέφερε άλλωστε και η κυρία ε, Σαργεντίνη η ερευνητική ας πούμε δημοσιογραφία είναι κάτι το πολύ θετικό και θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Θα ήθελα περισσότερες συστάσεις ε, για την ε, ε, ανάπτυξη της ειδησιογραφικής δημοσιογραφίας και της ερευνητική δημοσιογραφίας. Νομίζω ότι αυτού του είδους ε, η δημοσιογραφία ε, σε πολλές ε, περιπτώσεις περιορίζεται. Και το βλέπουμε πολύ και στις ίδιες τις Βρυξέλλες. μειώνεται ο αριθμός των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες ενώ η σημασία του, ε, των όσων συμβαίνουν εδώ αυξάνεται. Ε, βλέπουμε και επομένως άμεσα πως ε, η οικονομική κρίση χαμηλώνει το επίπεδο της δημοσιογραφίας, της πραγματικής δημοσιογραφίας. Σίγουρα λοιπόν και για αυτό το θέμα θα υποβάλω τροπολογίες. Αναφέρθηκα ήδη στον ε, νόμο του ανταγωνισμού. Αυτός είναι, αυτή είναι βασική προϋπόθεση για την ανεξαρτησία των ε, ε, της δημοσιογραφίας. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει καλή ισορροπία ανάμεσα στην εσωτερική αγορά αφενός και τις ιδιαίτερες πολιτιστικές παραδόσεις αφετέρου εάν ο ανταγωνισμός οδηγήσει ε, σε ε, επιφανειακή δημοσιογραφία και τα λοιπά, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να προσέξουμε. Βεβαίως, οι νόμοι του ανταγωνισμού έχουν επίσης ε, και άσχημες επιπτώσεις με τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά ε, τα κονδύλια, τα δημόσια κονδύλια που χρησιμοποιούνται για, την, ε, ε, που χρησιμοποιούνται για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Αλλά εδώ έχουμε περικοπές παντού, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικά τα δημόσια μέσα, αλλά ότι δεν έχουν χρήματα έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά. Τελικά, τελική μου παρουσίαση. αυτά που συνέβησαν στην ΙΚΟ και σχετική επιστολή στον Πρόεδρο ε, με προβληματίζουν. Έχουμε μία... Ε, εκεί υπάρχει μία, ένα κείμενο το οποίο ε, βάζει σε πολύ δύσκολη θέση τους δημοσιογράφους. Εάν δημοσιοποιήσουν δηλαδή στοιχεία ανταγωνισμού, στοιχεία για επιχειρήσεις και ε, και ε, ε, κερδίσει χρήματα η εφημερίδα από τη δημοσίευση αυτή, τότε μπορούν να υπάρξουν εναντίον της, της εφημερίδας ποινικέ διώξεις. Εδώ υπάρχει ε, σαν απόρρια μιας έκθεσης της ΕΚΟΝ ε, προσφυγή σε ε, ποινικό δίκαιο που όμως δεν έχει γίνει καλά και προετοιμασμένα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο το θέμα αυτό. Επίσης πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και νομίζω ότι θα πρέπει στην σύσταση, αυτή η σύσταση να αναφέρεται και στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ήλτσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη Ρενάτε Βέμπερ για την εξαιρετική της έκθεση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά θα, θα ακολουθήσουν πολλές ε, προτάσεις ε, τροπολογίας. Αυτό βέβαια αποδεικνύει πόσο σοβαρή είναι η έκθεση. Βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία, σε μία εποχή όπου το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης είναι κάτι το, το κοινό, που ακόμη και στις χώρες όπου υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα των, ε, ε, του τύπου, του γραπτού τύπου είναι καταστροφικό σε ορισμένες χώρες. Εκεί όπου το σύστημα διανομής αποφασίζουν το χρόνο ζωής σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα και αποφασίζουν πότε αυτή η εφημερίδα θα εξαφανιστεί από την αγορά. Είναι φανερό ότι η συγκέντρωση των ΜΜΕ οδηγεί και στην ε, συγκέντρωση της ε, διανομής. Για το θέμα των μίντια και της ε, διαφήμισης σύμφωνη, αλλά υπάρχει ένα, μια άλλη διασύνδεση, ΜΜΕ και πολιτικό περιβάλλον. Ορισμένα έψιλων είναι τα θύματα των, ε, των πόθων τους. Σε πολλές ε, χώρες ε, βλέπουμε ο τύπος να αισθάνεται μέρος του εκτελεστικού οργάνου. Βλέπουμε τον τύπο σε πολλές χώρες να μην είναι από τη μεριά των πολιτών, Ε, βλέπουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν υπέρ αυτών την αρχή της επικουρικότητας. Εμείς σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας. Και γι' αυτό δρούν με τρόπο μη δημοκρατικό. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε ένα profiling μεμονωμένο, αλλά ένα profiling συνολικό όλων των ιδιοκτητών εφημερίδων, όλων των ιδιοκτητών ΜΜΕ πρέπει να έχουμε ελάχιστα ζητούμενα. Ζητούμενα που δεν πρέπει να είναι σχολαστικά σχόλια, πρέπει να είναι προστακτικά σχόλια τα οποία θα μας βοηθήσουν. Εμείς Πρέπει να δούμε πώς δουλεύει η Europol, πώς δουλεύει η Frontex. Και να φτιάξουμε μια ομάδα, όπως είπε και η Ρενάτε, γιατί είμαστε τόσο περιοριστικοί Εμείς δεν πρέπει να δίνουμε ελευθερίες στα άτομα τα οποία επηρεάζουν τα μίντια. Πρέπει να τελειώσετε, να ολοκληρώσετε κυρία Βέμπερ, γιατί θα έρθει και ο κύριος Κοέγιο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στις 11 ξεκινάει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, λέει η κυρία Βέμπερ, για τα σχόλια που έκαναν. Δεν θέλω να απαντήσω διεξοδικά και εξαντλητικά σε όλα τα σχόλια γιατί δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι την 6η Νοεμβρίου έχουμε προβλέψει ε, ακρόαση. Η προθεσμία κατάθεση είναι η 8η Νοεμβρίου και επομένως θα ακούσουμε ε, τα θέματα της ακρόασης, ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε και μετά θα έχουμε ε, την δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογίες. Για μία ακόμα φορά πάντως να πρέπει, θέλω να τονίσω το εξής ακούστηκε ότι αν δεν υπάρχει νομοθεσία πρέπει να δημιουργήσουμε. Ίσως αυτό να είναι λίγο δύσκολο γιατί και επικίνδυνο γιατί μερικοί μπορούν να πούνε αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο κτλ. Έχουμε το άρθρο 11 της ε, ε, της χάρτας ε, σε συνεργασία με το άρθρο σε συνδυασμό συγγνώμη, με το άρθρο 2 της συνθήκης λειτουργίας νομίζω ότι αυτή η συνδυασμένη δυνατότητα μας δίνει δυνατότητα δράσης οποιαδήποτε στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταλάβαμε ότι η Κομισιόν δεν ήθελε σε αυτό το στάδιο να συμμετάσχει στη συζήτηση. Ε? Περιμένετε να δείτε τις τροπολογίες. Έτσι καταλάβαμε ότι δεν ήθελε η Κομισιόν να μιλήσει τώρα. Οπότε ε, να ευχαριστήσουμε την κυρία Βέμπερ για την παρουσίαση. Προτείνω να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, σημειώνοντας βέβαια ότι η ακρόαση ΛΥΜΠΕ θα οργανωθεί στα πλαίσια της έκθεσης αυτής ε, στις 6 Νοεμβρίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και η προθεσμία υποκατάθεση τροπολογιών είναι η 8 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ωραία. Και προχωρούμε στον κύριο Κοέγιο που θα μας μιλήσει για λίγο για το SIS, σύστημα ε, πληροφόρησης Schengen. Έχετε το λόγο κύριε Κοέγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε είχε προβλεφθεί ψηφοφορία στο θέμα αυτό, τη μετάβαση στο καινούριο δεύτερης γενιάς σύστημα πληροφοριών Schengen τώρα στις 11. Τι συνέβη όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε τρία πράγματα για τη μετάβαση. Πρώτον, χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν γιατί είναι πολύ καλύτερη ε, σχετικά με την ε, νομική βεβαιότητα, ασφάλεια, την ασφάλεια δικαίου. Δεύτερον, μπαίνουμε σε ταχεία διαδικασία για να επιτρέψουμε ε, στα κράτη-μέλη να ωφεληθούν από την γραμμή του προϋπολογισμού που υπάρχει φέτος για να στηρίξει τα μέτρα στα εθνικά συστήματα και τρίτον κάναμε, καταθέσαμε κάποιες τροπολογίες για την βελτίωση της προστασίας δεδομένων ε, στους φακέλους υπομετάβαση. Τι συνέβη τώρα. Το Συμβούλιο αποφάσισε να χωρίσει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από διαδικαστικής πλευράς δεν δουλεύουμε τώρα πάνω στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα έπρεπε να δουλέψουμε πάνω στις δύο νέες προτάσεις του Συμβουλίου. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να ψηφίσουμε σήμερα, όπως είχε προβλεφθεί, και πρέπει να αλλάξουμε τις τροπολογίες μας από την αρχική πρόταση να πάμε στα δύο καινούρια κείμενα που έχουμε και έχουν που κυκλοφόρησαν πριν από λίγα λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη συμβιβαστική λύση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ωφεληθούν φέτος από τη γραμμή του προϋπολογισμού, προτείνω να ακολουθήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στον κανόνα 46 του κανονισμού μας. Ε, έτσι θα επιταχύνουμε την διαδικασία, δεν πρόκειται να φτιάξουμε κάτι καινούριο, θα αλλάξουμε τις τροπολογίες που είχαμε ήδη ε, καταθέσει για το αρχικό πρωτότυπο κείμενο, να τις πάμε στο, στα καινούργια δύο καινούργια κείμενα έτσι θα μπορέσει η Επιτροπή Λίμπε να συμφωνήσει επί ενός κειμένου και να ψηφίσει σε μια συνεδρία στο Στρασβούργο κατά την ε, συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Αυτό προτείνω στους, ε, σε εσά, στους Κιώδης και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Λίμπε. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο. Ε, η Κομισιόν, η Κυπριακή Προεδρία θέλει να παρέμβει, θέλουν να παρέμβουν σχετικά με το θέμα αυτό της μετάβασης στο δεύτερο εις γενιά σύστημα SIS, η Προεδρία. Παρακαλώ, η Κυπριακή Προεδρία θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους σας. Η Προεδρία και το Συμβούλιο θα ήθελα να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για την εργασία που έχει εκπονήσει για το θέμα αυτό, αλλά και για την ευελιξία την οποία έχει δείξει στην συνεργασία που έδειξε για αυτήν την επιταχυμένη διαδικασία. Βεβαίως ε, αποδίδεται μεγάλη σημασία σε όλες τις προτινόμενες, θα δοθεί μεγάλη σημασία στις προτινόμενες τροπολογίες και θα ληφθούν όλες οι υπόψη. Θα ήθελα τέλος να πω ότι δεν παραβλέπουμε την σημασία του συστήματος ΣΥΣ ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε ε, στην αρχή του 2013, στο πρώτο τρίμηνο, να αρχίσει να λειτουργεί. Ε, ευχαριστούμε την Προεδρία. Η Κομισιόν δεν θέλει να πάρει το λόγο. No further comments. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ακούσαμε όλες τις υπεκυροποιημένες θέσεις όσον αφορά την έκθεση αυτή. για το σύστημα ΣΥΣ δεύτερης γενιάς, την αναδιατύπωση δηλαδή, να σας πω ότι ακούσαμε τον εισηγητή και την πρότασή του, δηλαδή να προχωρήσουμε στην απλοποιημένη διαδικασία βάσει του κανονισμού 46 και για τα δύο κείμενα του Συμβουλίου. Σύστημα πληροφοριών ΣΥΣ και τις δύο προτάσεις εάν συμφωνείτε όλοι, δηλαδή εννοώ εάν δεν αντιτίθεται κανείς στην πρόταση που υπέβαλε ο κύριος Κοέγιο τότε θεωρείται συμφωνηθήσα. Είναι σαφές αυτό. Συμφωνήσαμε λοιπόν και συμφωνείτε κι εσείς να χρησιμοποιήσουμε την απλουστευμένη διαδικασία βάσει του άρθρου 46. Άψογα ευχαριστούμε τον κύριο Κοέγιο για την έκθεσή του. Και περνάμε τώρα Μάλλον όχι. Ε, σταματάμε για λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μην λησμονήσετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ψηφοφορίες. Σε δύο-τρία λεπτάκια ξεκινάμε. Συνεχίζουμε. Κάποιες ψηφοφορίες έχουμε, κάποιες έχουν αναβληθεί, αλλά μας έμειναν και μερικές. Να προχωρήσουμε. Προχωρούμε. Η πρώτη πραγματική ψηφοφορία που θα έχουμε είναι επί του σχεδίου γνωμοδότησης για τις ρήτρες αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης, ε, πολιτικές και επιχειρησιακές διαστάσεις, ο κύριος Μπουσούτιλ. Ε, οι ρήτρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αμοιβαία άμυνα και αλληλεγγύη, πολιτικέ και επιχειρησιακέ διαστάσει. Προχωρούμε. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Όχι. Καταπίπτει η 5. Έχει καταπέσει. Α, ως προσθήκη. Την 5 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 6, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 7, υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 8, υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος, γιατί βλέπω εδώ κάποια ε, διαφοροποίηση, αλλά θέλω να ξέρω ποιοι ακριβώς είναι υπέρ και ποιοι ακριβώς είναι κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της 17. Πέρας. «21 υπέρ, 17 κατά, 18 ε, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όσο τροποποιηθεί. Πάμε για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Και τι έχουμε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έκλεισε η ψηφοφορία. Α, πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Ε, δεν λειτουργήσε το μηχάνημα. Για να ξαναδοκιμάσουμε. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Μάλιστα, 33 υπέρ, 3 κατά με 4 αποχές. Μπράβο, κύριε Μπουσουτήλ, αξίζεται συγχαρητήρια μετά από το αποτέλεσμα αυτό. Και προχωρούμε τώρα. Υπάρχει δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Τώρα πάμε στην ε, ψηφοφορία. Σχέδιο γνωμοδότηση για την πρόταση του για κανονισμό Συμβουλίου για Ευρώπη των ε, Πολιτών. Ένα πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020. Πάμε στην τροπολογία 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτό. 39. Υπέρ κατά αποχές δεκτή, 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 41 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 42 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, πέντε, υπέρ. Όχι, συγγνώμη, τέσσερα Προσπέρασα μία, λέει ο πρόεδρος, στην τροπολογία τέσσερα Αυτή θα ψηφίσουμε τώρα. Πάμε πίσω λοιπόν στην τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 5 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 6, υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ. Α, όχι, συγγνώμη, 43. Θα ψηφίσουμε 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 θέλετε να ελέγξουμε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στην 10 μάλιστα ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία τροπολογία 10 πέρας Mm. Πρόβλημα. Από απερίφθη 18 υπέρ 23 κατά. Ψηφίζουμε τις 44 λοιπόν. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ όχι πια αυτή η 11 υπέρ την 11 ψηφίζουμε 45 κατέπεσε κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά, αποχές δεκτή, 18 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 51 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 19 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 20 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 52 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εννοώ το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ 56 την 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ ε, κατά αποχές δεκτή τώρα λογική σκέψεις και αναφορικές προτάσεις 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές απο... Ε, ε, εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ 36 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζομαι το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τώρα Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 40 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Ε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σόγκορ. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες νομίζω. Και τώρα Πάμε στην Frontex. Λοιπόν, να δώσουμε λίγα λεπτά για να φύγουν όσοι θέλουν σιωπηλά για να, και να καλωσορίσουμε τον διευθυντή του Frontex, τον κύριο Ιλκα Λάιτινεν, σε ένα λεπτό. Please, colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. People willing to leave the room, do it please in silence from now on. Those of you in the room. Λοιπόν, δώσαμε λίγα λεπτά έτσι ώστε να εγκαταλείψουν ησύχως όσοι θέλουν την αίθουσα, να σταματήσουν τα πηγαδάκια και οι διμερείς έτσι κουβεντούλες, γιατί είμαστε εδώ για να ακούσουμε τον, ε, τον ε, προσκεκλημένο μας κύριος, κύριο Ικα Λατίνεν ο οποίος είναι διευθυντής της υπηρεσίας Frontex και ο οποίος ε, είναι εδώ για να μας κάνει μια παρουσίαση. Μετά το πέρας παρουσίαση του κυρίου Λαϊτίνεν θα έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Να θυμίσουμε πάντως ότι εγκρίναμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τροποποίηση του προϋπολογισμού της Frontex 2013 βάζοντας σε αποθεματικό περίπου 10 ε, εκατομμύρια μέχρι ότου ο Διευθυντής κ. Λαϊτίνεν παρουσιάσει εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα αναλάβει η ε, Frontex έτσι ώστε να βελτιώσει τα, μέσα, ε, τα μέτρα θαλάσσιας διάθεσης μεταναστών και να συμπεριληφθεί αυτό στην νέα εντολή του Frontex.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 Ε, μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που για μία ακόμα φορά βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έτσι ώστε να σας κάνω μια αναφορά σχετικά με τα πρακτικά βήματα τα οποία έχει αναλάβει η υπηρεσία Frontex έτσι ώστε ε, να διασώζει ζωές στην θάλασσα. Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα αυτό εξ αρχής. Επιτρέψτε μου πάντως να ξεκινήσω με μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα αυτό. Από τον Αύγουστο τρέχοντος έτους ε, έχουμε ε, δει ε, μεγάλη μετατόπιση του κέντρου βάρους των δραστηριοτήτων τα, τον προηγούμενο καιρό τα μεγαλύτερα ποσοστά τα βλέπαμε στα χερσαία σύνορα, ενώ τώρα ξαναφτάσαμε στα θαλάσσια σύνορα. Το βάρος ξαναέχει πέσει στα θαλάσσια σύνορα. Σε γενικές γραμμές πάντως τα θαλάσσια σύνορα, η θάλασσα γενικότερα ε, φαίνεται να ε, αντιμετωπίζει μεγαλύτερο βάρος και επομένως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτημα ε, της συζήτησης των πρακτικών μέσων για τη βελτίωση των μέτρων θαλάσσιας διάσωσης. Το δεύτερο σημείο που θα αναφέρω είναι η ατομική μεμονωμένη προσέγγιση για την εργασία και τον ρόλο που παίζουν οι ακτοφυλακές στην διάσωση ανθρωπίνων ζώων. Όταν ε, οι καταστάσεις ε, είναι καλές, ε, βεβαίως δεν συμβαίνουν προβλήματα, αλλά οι συνθήκες μέσα στις οποίες προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπινες ζωές και οι επιχειρήσεις διάσωσης αξίζουν το σεβασμό όλων. Το τρίτο μου σημείο θα αφορά τις αρμοδιότητες που η Frontex και τα κράτη-μέλη έχουν κατά την έννοια των θεμάτων που μας απασχολούν. Έχουμε καλή ισορροπία και ομαδική προσέγγιση, πνεύμα ομαδικής προσέγγισης όσον αφορά τις αρμοδιότητες αυτές. Υπάρχει μία πρόκληση σε σχέση με τον συντονισμό ε, και την οργάνωση κοινών, ε, ε, κοινών επιχειρήσεων διάσωσης στη θάλασσα. Σε πολλές χώρες μέλη το κέντρο συντονισμού των θαλασσίων διασώσεων δεν είναι η ίδια αρχή ε, που ασχολείται με τις κοινέ επιχειρήσεις ε, διάσωσης υπό την Frontex. Αυτό βεβαίως δυσκολεύει την κατάσταση και εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε πρακτικά μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός. Βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί απανταχούει στον κόσμο όσον αφορά ε, τις ε, επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης, μπορούμε να βρούμε διάφορες ε, κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία των unsafe boats, ανασφαλών μη ασφαλών σκαφών. 90% των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο στην κατηγορία αυτή έλαβαν χώρα ε, υπό την κοινή ε, διαχείριση της ε, Frontex στην οποία συμμετείχαν οι δυνάμεις της Frontex έμεσα ή άμεσα. 90% των ατυχημάτων των μη ασφαλών σκαφών λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια των κοινών επιχειρήσεων της Frontex. Θα σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία του 2011 καταγράψαμε 246 ε, υποθέσεις ανείχνευσης και διάσωσης, όπου παραπάνω από 23.000 ε, άνθρωποι διασώθησαν. 246 υποθέσεις με 23.000 και πλέον διασωθέντες. Φέτος ο αριθμός των υποθέσεων έχει φτάσει μέχρι τώρα τις 118. Ε, με ε, διασωθέντες λίγο λιγότερους από 40.000. Ε, είναι ε, σαφής επομένως η βελτίωση της κατάστασης λιγότερες υποθέσεις με περισσότερους διασωθέντες. Μία άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση προς το ζήτημα αυτό είναι η σύγκριση ανάμεσα στην ανείχνευση λαθρομεταναστών πόσοι από αυτούς διασώθησαν στη θάλασσα θάλασσα. 38 ε, ήταν το, το ποσοστό το 2011. Αυτό σημαίνει ότι 4 στους 10 περίπου λάθρομετανάστες βρίσκονται ε, ε, σε συνθήκες επικίνδυνες στην θάλασσα. Φέτος το ποσοστό έχει φτάσει στο 33%. Γιατί το αναφέρω αυτό με τέτοια λεπτομέρεια. Μα γιατί αυτό αποτελεί και την ε, αιτιολόγηση ότι σημείο κίνησης ε, για την διαχείριση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των ε, θαλασσίων επιχειρήσεων είναι ότι οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσουμε οι περιπτώσεις θαλάσσιας διάσωσης. Αυτό είναι σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των εν λόγω δραστηριοτήτων. Μου ζητήσατε να αναφερθώ στα πρακτικά βήματα, γι' αυτό λοιπόν θα ασχοληθώ με συγκεκριμένα πράγματα, τι έχουμε κάνει δηλαδή όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διαχείριση. Πρώτον, πρέπει να ε, ορίσουμε την ε, περιοχή της ε, επέμβασης. Υπάρχουν, θα πρέπει να καθοριστεί λοιπόν η επιχειρησιακή περιοχή γιατί και να γίνει η ανάλυση κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι ένας σημαντικός παράγων ε, που μας λέει που θα λάβει χώρα η επιχείρηση είναι η δυνατότητα να σώσουμε ε, ανθρώπινες ζωές. Το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη διαδικασία ε, προετοιμασίας και σχεδιασμού βλέπουμε τις παλαιές στατιστικές. Ε, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος, η καλύτερη στιγμή για να αναλυφθεί δράση. Οι προετοιμασίες ε, για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σχηδείς. Το σχέδιο είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικό. Ε, εκεί όμως συνυπολογίζονται και οι δυνάμεις επιτόπου και οι ε, συμμετέχουσες ε, χώρες οι οποίες θα πρέπει να επικυρώσουν το σχεδιασμό. Έχουμε μια σταθερή ρήτρα όσον αφορά τις οδηγίες που δίνουμε ε, εμείς αναπτύξαμε αυτές τις κοινέ οδηγίες στη διάρκεια της ε, πολυετούς δραστηριότητας της Frontex και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα ικανό σημείο λεπτομερίας καθώς επίσης και ε, σε ένα ικανό σημείο ακρίβειας όσον αφορά την αντίδραση σε κάθε περιστατικό. Επίσης πρέπει να καθοριστούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του κάθε συμμετέχοντος. Όπως είπα υπάρχει διαφορά ε, ε, ανάμεσα, πολύ συχνά ανάμεσα στο Εθνικό ε, Κέντρο Θαλάσσιου Συντονισμού και το κέντρο το οποίο συντονίζει σε συνεργασία με την Frontex. Σε μερικές περιπτώσεις ε, πρέπει να γίνει μετατόπιση έτσι ώστε να υπάρχει ένας φορέας. Αυτή η μετατόπιση, αυτή η μετάβαση θα γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται. Η εξάσκηση είναι ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο σχετικά με τις θαλάσσιες ε, επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρξει εξάσκηση όσον αφορά την συνεργασία και το συντονισμό με τα εθνικά κέντρα και τα διεθνή ε, κέντρα ε, ε, θαλάσσιας συνεργασίας και να αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε μονάχα την μονότονη περιπολία των σκαφών. Διαρκώς εξασκούμε τα πληρώματα, διαρκώς αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες καταστάσεις ένα πολύ σημαντικό σκέλος, το οποίο επίσης αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, είναι η υποχρέωση πληροφόρησης ε, του Κέντρου Συντονισμού των Θαλασσίων Διασώσεων σχετικά με τα μέσα τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση ε, Frontex, δηλαδή πότε περιπολούν, πού και με ποια μέσα. Ε, έτσι ώστε η ε, Frontex να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή σε ποια περιοχή μπορεί να αναπτύξει ποιες και πόσες δυνάμεις σε μια περίπτωση θαλάσσιας διάσωσης. Αυτά όσον αφορά το δεύτερο ε, σκέλος. Το τρίτο σκέλος αφορά τον εξοπλισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινούμε τον σχεδιασμό και τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη να γνωρίζουμε ε, τι εξοπλισμό θα έχουν, τι ικανότητα θα έχουν για συμμετοχή και εμπλοκή σε θαλάσσιες διασώσεις. Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι τα σκάφη, μπορεί να είναι τα εναέρια μέσα, έτσι ώστε να... και ο βασικός εξοπλισμός ανείχνευσης. Έχουμε επίσης ε, ε, και μία ε, πλήρη εποπτεία όλων των εξοπλισμών και όλων των μέσων παρακολούθησης. Επίσης σημαντικό σημείο είναι η ετοιμότητα ε, κυρίως των σκαφών ε, να εμπλακούν σε θαλάσσιες διασώσεις. Ε, βεβαίως έχουμε και συγκεκριμένες προβλέψεις όσον αφορά τον αριθμό των προμηθειών, το εύρος των προμηθειών, νερό, τροφή, νερό, εξοπλισμός, κουβέρτες κτλ. Γίνεται λοιπόν ένα pre-screening όλων των εξοπλισμών, του τύπου σκαφών, των εναερίων μέσων κτλ. Το επόμενο πρακτικό μου βήμα αφορά την ε, ε, εξάσκηση. Έχουμε αναπτύξει ε, κάποια μαθήματα πρακτικά όσον αφορά τις θαλάσσιες διασώσεις και οι ασκήσεις αυτές αφορούν τα σκάφη, τα εναέρια μέσα και το προσωπικό τους. Ε, είναι σημαντικό ε, όλοι, όλα τα μέλη, όλα τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν σε θαλάσσιες διασώσεις να έχουν προσωπικό και μέσα τα οποία θα έχουν περάσει από την απαραίτητη εξάσκηση και βασιζόμαστε εδώ στα πρότυπα του IMO, του Διεθνούς ε, Θαλασσίου Οργανισμού. Αυτά είναι τα πρακτικά βήματα τα οποία αναλαμβάνουμε έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις έτσι ώστε και τα μέσα και ο εξοπλισμός αλλά και τα άτομα να είναι καλά προετοιμασμένα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ε, στα κατά κάποιο τρόπο δευτερεύοντα μέτρα τα οποία θα πρέπει να θεωρηθούν και αυτά πρακτικά βήματα. Πρώτα θα αναφερθώ στην διυπηρεσιακή συνεργασία. Έχουμε εδώ λοιπόν την Frontex, την Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας, την Υπηρεσία Ελέγχου των Αλλιευμάτων, ε, την ε, Υπηρεσία Στήριξης ε, του Ασύλου, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Κέντρο. Όλοι αυτοί πρέπει να συνεργάζονται ε, αλλά με μερικές υπηρεσίες ε, για τον με αυτήν του ελέγχου των αλλιευμάτων ε, και της θαλάσσιας ασφάλειας έχουμε προχωρήσει σε κοινέ διαδικασίες και επιχειρήσεις κυρίως στα ισπανικά ύδατα. Εμείς θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Είναι ένας ε, όρος που πλέον εμφανίζεται ως πυρηνικός όσον αφορά ε, το θέμα της θαλάσσιας διάσωσης. Η διάσωση ανθρωπίνων ζώων συνδέεται άμεσα με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πω δύο λόγια για την στρατηγική της υπηρεσίας μας όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μη λησμονώντας βεβαίως και τη συζήτηση που είχαμε ε, πριν ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τα θέματα αυτά. Είμαι ευτυχής διότι μπορώ να σας πω ότι ε, ο υπεύθυνος ε, για θεμελιώδη δικαιώματα της υπηρεσίας έχει οριστεί πλέον. Ε, είναι γυναίκα και μας και κοινοποίησε στην Frontex ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τα καθήκοντά της άμεσα. Δεύτερον, όσον αφορά την Συμβουλευτική Επιτροπή, είναι γεγονός ότι είχαμε την πρώτη συνάντηση την 15η Σεπτεμβρίου και την πρώτη επίσημη συνάντηση ε, την 16η Οκτωβρίου. Θα λάβει η χώρα λοιπόν η πρώτη, αυτή ήταν η ανεπίσημη του Σεπτεμβρίου. Η επίσημη θα λάβει η χώρα την 16η Οκτωβρίου και βεβαίως καλό τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να παραστεί σε αυτήν την πρώτη ε, ε, συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιθεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνεργάζεται άμεσα με την Frontex. Χθες όλο το πρωί ε, συζήτησα επί μακρόν με τον ε, συνάδελφό μου της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γιατί η διάσωση ανθρωπίνων ζώων είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τους δυο μας. Έχει γίνει πολλή δουλειά, η συνεργασία όμως έχει καρποφορήσει. Κύριε Πρόεδρε, τελικό μου σημείο θα είναι η Eurosur. δεν είναι απλώς ωραία λόγια όταν μιλάμε για τη Eurozone. Πρόκειται για ενδυνάμωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εντός συνόλου της να σώσει ανθρώπινες ζωές. Ε, ε, χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο τα αναλυτικά εργαλεία, τα σωστικά εργαλεία, ε, έχουμε μία πληρέστερη εικόνα έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε την ικανότητα διάσωσης ανθρωπίνων ζώων. Υπάρχουν και κάποια παρεμπίπτοντα ζητήματα τα οποία έχει αναπτύξει η Frontex και που θα ενταχθούν αργότερα στη Eurosur. Πρώτον, η θέση της ε, Frontex στο σύστημα ε, σημαίνει ότι έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ε, βάσει του οποίου μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ακριβή θέση όλων των ε, συμμετεχόντων ε, μονάδων έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να τις αναπτύξουμε όσο γίνεται γρηγορότερα εάν παραστεί ανάγκη θαλάσσιας διάσωσης. Πολύ σημαντικός παράγων επίσης ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα ενσωματώσουμε δηλαδή ε, να, κάνουμε μια, να αναπτύξουμε συμβατή εικόνα. Δηλαδή στο μέλλον θα έχουμε την δυνατότητα επιγραμμικής ε, ανταλλαγής εικόνας ε, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται άμεσα σε διαδικασίες διάσωσης και φυσικά αυτό θα αναπτύξει, θα μεγαλώσει την σωστική ικανότητα που έχουμε. Summing uh, Ολοκληρώνοντας, ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε αναλάβει πολλά πρακτικά βήματα ε, και πολλά τα οποία θα, ε, κάνουμε στο μέλλον. Το να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιχείρηση θαλάσσιας διάσωσης δεν αποτελεί εξαίρεση ή ιδιαίτερη στιγμή των επιχειρήσεών μας. Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ε, ε, το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πάντα οι ίδιοι με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την συνεργασία με τη Frontex σημαίνει ότι πρέπει σιγά σιγά ε, να ταυτιστούν οι υπηρεσίες έτσι ώστε η συνεργασία να είναι πιο, πιο άμεση και πιο γρήγορη. Επίσης θα πρέπει να ταυτιστεί η ορισμός για την ε, κατάσταση κινδύνου. Σε ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, δεν έχουν τον ίδιο ορισμό για την κατάσταση κινδύνου στην θάλασσα όλες οι χώρες. Θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα να πω δύο λόγια για το 2013. Θυμηθείτε τι σας είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ε, πλέον στην θάλασσα έχει πέσει το κέντρο ε, βάρους. Η κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως γνωρίζετε, ε, είναι άγνωστη για την ώρα. Και η υπηρεσία θέλει να είναι έτοιμη ε, για ε, θαλάσσιες ε, επιχειρήσεις, οι οποίες όμως είναι και οι πιο ακριβές επιχειρήσεις, διότι χρειάζεται πολλαπλός εξοπλισμός και ένα αέρια μέσα και σκάφη κτλ. Είναι δύσκολο για μας να προετοιμάσουμε τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας, εάν δεν γνωρίζουμε τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά ήθελα να σας πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να σας μιλήσω για αυτά τα πρακτικά βήματα που αναλαμβάνει η Frontex έτσι ώστε να βελτιώσει την, ε, ε τις επιχειρήσεις θαλάσσιας, θαλάσσιας διάσωσης και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαϊτίνα. Να αρχίζει η συζήτηση. Ο κύριος Παπα-Νικολάου ζητεί πρώτος το λόγο. Mr. Chairman, not the first. Οι συντονιστέ ε, δεν πρέπει να λάβουν πρώτοι το λόγο. Βέβαια, να ζητήσουν το λόγο και έχουν προτεραιότητα όταν θελήσουν να παρέμβουν στη συζήτηση. Αν έχει όμως, εσείς θα πάρετε το λόγο. Κύριε Μπουσούτιλ, δεν είστε υποχρεωμένος. Θέλετε να μιλήσετε πρώτος. Ε, είναι και θέμα περηφάνειας. Ε, ε δεν είναι θέμα περηφάνειας για να ποιο θα πάρει πρώτος το λόγο. Δεν θα το δούμε ανταγωνιστικά, ούτε εγώ θα το δω ανταγωνιστικά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λάιτινεν που ήρθε εδώ, λέει ο κύριο Μπουσουτήλ. Πάντα λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επαφή μαζί σας και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται επίτόπου. επί τόπου ώστε να γνωρίζουμε τις επιχειρήσεις του οργανισμού. Άλλωστε αποδίδει η Επιτροπή μας μεγάλη σημασία στο ρόλο σας. Καταρχήν εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου, διότι ο υπεύθυνος, ε, ε, έχει οριστεί κάποιος υπεύθυνος για τα ανθρώπινα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα υπάρχει αυτό στην ενημερωμένη νομοθεσία και πολύ χαίρομαι που ανέλαβε θα αναλάβει καθήκοντα σύντομα στα μέσα Δεκεμβρίου όπως μας είπατε. Ωραία, ως προς αυτό λοιπόν. Τώρα, το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα. Προφανώς και χρειάζεστε και εξοπλισμό για να είστε βέβαιοι ότι το ευαίσθητο αυτό θέμα θα αντιμετωπίζεται όπως πρέπει. Δεν έχει να κάνει με την προθυμία να σωθούν ζωές στη θάλασσα. Πρέπει να φροντίζομαι ότι υπάρχουν και τα απαραίτητα κεφάλαια υποδομή αλλά και εκπαίδευση, κατάρτιση. Την αναφέρατε εσείς την εκπαίδευση, κατάρτιση και αυτό είναι καλό. Και όταν επισκεφθήκαμε στη Βαρσοβία τα γραφεία σας μας έδειξαν τη βίβλο της ε, του, προγράμματος, ε, του, του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευση. Αλλά τι γίνεται με την υποδομή. Έχετε τη δυνατότητα να μισθώσετε ή να αγοράσετε ε, περιουσιακά στοιχεία. Κάποια στοιχεία μπορούν να αγοραστούν ή να μισθωθούν λοιπόν και γι' αυτό το σκοπό. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θέσω αν μπορώ αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της Frontex που επίσης συνδέονται άρρηκτα με το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα. Ξέρετε κύριε Λάιτινεν ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα θεωρούνται άκυρες αν και ακόμα ενισχύει μέχρι ότου αλλάξουν και εμείς περιμένουμε τώρα την αντίδραση της Κομισιόν στις εξελίξεις αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω, στην πράξη αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιήθηκαν καθόλου την προηγούμενη διετία, ακολουθήθηκαν και στο φως της απόφασης του δικαστηρίου ο οργανισμός Frontex έχει αναφερθεί στην Κομισιόν για να πει πώς θα αλλάξουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και αν έγινε αυτό ε, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε και μας όπως ενημερώσατε την Κομισιόν. Ευχαριστώ η κυρία Γκυγιόμ και μετά ο κύριος Παπα-Νικολάου. Mm είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλες τις πολιτικές ομάδες και μετά ο κύριος Παπα-Νικολάου. Συγγνώμη Γιώργο, δεν είμαι συντονίστρια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Εσείς αναφέρατε στην, ε, το θέμα της ε, πιθανότητας. Είναι περίεργο να ακούει κανείς ε, αυτήν την αρχή ε, της ε, πιθανότητας διότι με τα, τις διάφορες επιχειρήσεις και τα διάφορα ε, κλεισίματα συνόρων οι διάφορες ε, πιθανότητες έχουν περιοριστεί. Πώς, μπορείτε, πώς εργάζεστε εσείς βάσει του νόμου των πιθανοτήτων και τα τελευταία χρόνια διαπιστώσατε αν υπάρχει σύμπτωση μεταξύ πιθανότητων και των επιχειρήσεων της Frontex. Τώρα και αυτό που έλεγε και ο Σάιμον ε, για τον ε, αξιωματούχο για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, σχετικά με το γενικό πλαίσιο το οποίο είχαμε συζητήσει κατά τη μεταρρύθμιση του Frontex. Θέλω να ξέρω Έχετε προχωρήσει ως προς την λειτουργικότητα αυτής της θέσης και για το θέμα της θαλάσσιας διάσωσης ε, θα ενταχθεί ε, στις αρμοδιότητες αυτού του αξιωματούχου, δηλαδή θα έχουμε έναν τέτοιο αξιωματούχο στο πλοίο, η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες πρακτικές, κάποιες γενικές ερωτήσεις έχω. Αρχίζω με τις πρακτικές. Μιλήσατε για ανάλυση κινδύνου, επικινδυνότητας που λαμβάνετε υπόψη ε, όταν υπάρχουν αποστολές διάσωσης ταυτόχρονα που θα γίνουν, πώς θα οργανωθούν. Αυτό δεν εκπλήσει γιατί αν είναι πολλοί μετανάστες θα είναι και πολλές οι ε, καταστάσεις διάσωσης, θα υπάρχουν προβλήματα στους ανθρώπους και εσείς πρέπει να πάτε εκεί για να αντιμετωπίσετε την ε, είσοδο ο χειμώνας και φαντάζομαι η εποχή που θα έχει πολλές θύελες στη θάλασσα κλπ. Ε, είναι η πιο δύσκολη περίοδος. Έρχονται όμως το καλοκαίρι περισσότεροι μετανάστες. Εσείς ε, πώς θα ενισχύσετε τις, επιχειρήσει επιχειρήσεις σας ε, για να λάβετε υπόψη σας τα προβλήματα διάσωσης του χειμώνα. Επίσης, πώς γίνεται ακριβώς η διάσωση, δηλαδή τι βήματα ακολουθείτε, πώς αντιμετωπίζετε τα σκάφη που έχουν πρόβλημα, πώς γίνεται πρακτικά αυτό. Επίσης μιλήσατε για πολλούς που σώσατε από προβλήματα στη θάλασσα. Και μετά αφού τους σώσετε, τι τους κάνετε, πού τους πάτε, τους ρωτάτε αν ε, θέλουν να ζητήσουν διεθνή προστασία, τι γίνεται με, τα, με αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, πιο γενικά θέματα. Όπως και ο Σάιμον χαίρομαι γιατί ο υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα θα αναλάβει τα δικαιώματά του. Του πήρε χρόνο, ε, άργησε πολύ. Θα χρειαστεί μια ισχυρή φωνή που να είναι και ορατή και να ακούγεται στον οργανισμό και να ακούγεται για τις αποφάσεις σας. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρακτικά πράγματα υπόψη μας, να τα χρησιμοποιούμε ως μέτρο μέτρησης, τι θα ισχύσει κάθε φορά για τη διάσωση. Παλιά ξέραμε που είναι κάποιος Αλλά το να ξέρει κανείς που είναι δεν λύνει πάντα το πρόβλημα, γιατί είχαμε 63 μετανάστες που είχαν πρόβλημα. 63 ε, πέθαναν, πάνω από 70 ήταν. Όλοι ήξεραν ε, που ήταν, τους είχαν δει τα σκάφη και τα ελικόπτερα, αλλά κανείς δεν πήγε να τους σώσει. Και 63 από αυτούς πέθαναν Εννέα μόνο νομίζω επιβίωσαν. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα της Frontex, από ό,τι γνωρίζω δεν υπήρχε συμμετοχή της άλλωστε, αλλά δείχνει αυτό ότι το να ξέρει κανείς που βρίσκονται οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα δεν σημαίνει ότι θα σωθούν, πρέπει να υπάρχει η προθυμία να τους σώσεις. Βέβαια αν υπάρχουν προβλήματα ε, που μπαίνει ο νόμος για να κυνηγήσει ε, αυτούς τους ανθρώπους όπως στην Ιταλία, περιπλέκονται τα πράγματα. Πάντως ε, είναι καλό που βλέπουμε ότι ασχολείστε τόσο πολύ με τις επιχειρήσεις διάσωσης. Βεβαίως, και δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι η Frontex είναι ο καλύτερο εξοπλισμένος οργανισμός για τη διάσωση. Γιατί βέβαια η Frontex είναι ε, ένας οργανισμός ελέγχου συνόρων. Δεν είναι οργανισμός διάσωσης, ούτε οργανισμός ασύλου, ούτε οργανισμός μετανάστευσης. Και ε, πολύ μετανάστες, μετανάστες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την επαφή συνοριοφυλάκων κάθε είδους. Επίσης, ε, τώρα ακολουθούν πιο μακρές και επίπονες ε, οδούς για να έρθουν. Είδαμε πώς μετατίθενται οι οδοί των μεταναστών που είναι πιο μακρές, πιο ε, επίπονοι, καλύπτουν περισσότερα θαλάσσια κομμάτια. Και το θεμελιώδες ερώτημα εδώ είναι αν ε, είναι ο καλύτερος οργανισμός σας για τη διάσωση ή αν δεν έχει νόημα. Έχουμε ακτοφυλακή, την ακτοφυλακή που είναι υπεύθυνη για αυτά. Δεν είναι πράγματα που αφορούν την, τον Οργανισμό Ελέγχου Συνόρων, που είναι η αποτροπή εισόδου. Γίνονται όμως διασώσεις. Οπότε υπάρχει αυτό το θέμα. Αν η διάσωση όμως πιάνει, καλύπτει τόσο σημαντικό κομμάτι της αποστολής και της δουλειάς σας, και αυτό ίσως είναι ερώτηση προς την Κομισιόν που εκπροσωπείται εδώ, δεν είναι καλή ιδέα να ε, αναθεωρήσουμε την εντολή άλλη μια φορά με, βάζοντας μεγαλύτερη εστίαση στο θέμα διάσωσης και να μεταφέρομαι ε, περισσότερα καθήκοντα της Frontex στο τομέα της διάσωσης για να προσπα... παρά να αποφασίσουμε ή παράλληλα με την αποτροπή εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Ρίσμπεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κίνεν για την ε, παρουσίασή του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθένα, δηλαδή το, τι ποιος κάνει τι, ποιες είναι οι διάφορες προθεσμίες, μας τα είπατε όλα αυτά. Επίσης, ε, ε, ικανοποιήθηκα ακούγοντας αυτές τις αναφορές όλη αυτή τη συζήτηση αυτή τη συζήτηση για τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν σήμερα την Ευρώπη μας όπως επίσης άκουσα με ευχαρίστηση το ότι η αξιωματούχος για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι γυναίκα. Τώρα για αυτήν την ιδέα των πιθανοτήτων και για τον καθορισμό της ζώνης επιχειρήσεων, αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα θέματα. Εμείς το είδαμε κατά την Αραβική Άνοιξη εκατοντάδες ε, χιλιάδες άτομα να θέλουν να, ε, διαφεύγουν από τη, από τη βία της Λιβύης στη Λιβύη και να μεταναστεύουν μαζικά. Να έρχονται δηλαδή προς τις ε, προς τις ευρωπαϊκές ακτές της Ευρώπης, τα εξωτερικά μας σύνορα. Εμείς ε, σήμερα και αρκετά ε, άπραγοι να αντιδράσουμε οι Ευρωπαίοι, βλέπουμε αυτή τη σφαγή στη Συρία. Ε, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος και με ποιον τρόπο. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι 230.000 Σύριοι έχουν πήγε από τη Συρία και μιλήσατε για ορισμένους που προσπάθησαν να διαφύγουν διαθαλάσσεις, εσείς όμως μιλήσατε και για την προετοίμαση, ε, σχεδιασμό Άρα φαντάζομαι έχετε μία ιδέα για το πώς θα βοηθήσουμε εμείς αυτούς τους ε, μελλοντικούς ε, πρόσφυγες οι οποίοι θα μπαρκάρουν κάποια στιγμή προς την Ευρώπη. Και ποιες ε, διατάξεις, τι μέτρα θα πάρει η Ευρώπη, τι θέση θα πάρει η Ευρώπη για τους ετούντες άσυλο που θα αρχίσουν να μας παρουσιάζονται σε λίγο. Και σχετικά με το ερώτημα ενός συναδέλφου, πού προβλέπετε να πάτε όλον αυτόν τον κόσμο τον οποίο θα, θα διασώσετε για να απαντήσετε συμπερασματικά δηλαδή ε, στο ποιο θα είναι πώς θα σεβαστείτε τις ανθρώπινες ζωές μαζί με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κύριε Στρενταφυλλίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Λάιτινεν και την ευκαιρία να μας μιλήσει για τη Frontex. Περιμένω και εγώ τις απαντήσεις στο σχόλιο του κυρίου Μπουσουτήλ για τις κατευθυντήριες γραμμές και την αλλαγή που πρέπει να λάβει η χώρα και αν εκλήθη Κομισιόν να κάνει κάτι εδώ. Θέλω συγκεκριμένα να ρωτήσω κάτι για τις επιχειρήσεις σας κάποιες επιχειρήσεις διάσωσης και αν αναχαιτίζεται τα σκάφη στη θάλασσα, γιατί εγώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα με τις δυνάμεις που μετέχουν στη Μάλτα σε επιχειρήσεις διάσωσης και δεν ε, αναχαιτίζουν γιατί δεν τους επιτρέπει ο νόμος. Λειτουργούν μόνο ε, στα θέματα έρευνας και διάσωσης. Εκεί μόνο επιχειρούν. Και όπως ο προηγούμενος ομιλητής θέλω να ξέρω τι κάνετε τους ανθρώπους που τους σώζετε. Είπατε ότι αρκετές χιλιάδες ήταν αυτοί που διεσώθησαν τους τελευταίους μήνες. Τους ε, επιβιβάζετε στο σκάφος και τους κάνετε έλεγχο ή τους ξαναγυρίζετε στην χώρα τους. Τι κάνετε. Και ε, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Κέλλερ προηγουμένως ε, σχετικά με τις αρμοδιότητες του οργανισμού υπήρξαν περιπτώσεις συγκρούσεις αρμοδιοτήτων που μπορεί να καθυστέρησαν τις επιχειρήσεις σας σε βάρος των επιχειρήσεων διάσωσης και αυτό δηλαδή να απέβει σε βάρος της διάσωσης. Ευχαριστώ η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να διευκρινίσω κάτι που αναφέρατε, ότι δεν υπάρχει σαφήνεια στον προϋπολογισμό της Frontex για το 2013. Δεν, θα, δεν αναμένονται περικοπές, οπότε είναι σαφές. Γιατί εσείς νιώθετε αυτή την ανασφάλεια, αν και ακόμα την έχει τελειώσει ο ε, δεύτερον, ε, άκουσα και αυτά που είπατε και κατάλαβα ότι υπάρχει διαφορά στην εντολή της Frontex σε σχέση με αυτά που είχα εγώ υπόψη μου. Διάσωση ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ευγενική εντολή, αλλά πάντα είχα την εντύπωση ότι η Frontex φυλάει τα σύνορα και ότι είχατε δυσκολία να σώζετε για ανθρώπους. Έτσι νόμιζα. Μπορείτε να μας πείτε τι δεν πήγε καλά στα συστήματα έρευνας και διάσωσης τον τελευταίο χρόνο, γιατί στη Μεσόγειο την περασμένη φορά, ε, τον περασμένο χρόνο πνίγηκαν κατά προσέγγιση 1500 και είδαμε συγκεκριμένα την έρευνα που έκανε το Συμβούλιο της Ευρώπης για το σκάφος με τους ανθρώπους που έφυγε από τη Λιβύη και έπλεε δύο εβδομάδες στη Μεσόγειο και όλοι ήξεραν πού ήταν το σκάφος, υπήρχε και ελικόπτερο που πετούσε από πάνω ενώ κανείς δεν τους διέσωσε και κάποια στιγμή ξαναγύρισαν ε, πίσω στην ξηρά και πέθαναν σχεδόν όλοι. Αυτά τα πράγματα πρέπει ειλικρινά να μας κάνουν να ντρεπόμαστε. Θέλω λοιπόν να δείτε λίγο αυτή τη δήλωσή σας ε ότι είσαστε εκεί για να σώζετε ανθρώπους, αφού εμείς βλέπουμε ανθρώπους να πνίγονται ακόμα και όταν μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είμαι ο τελευταίος, αλλά είναι καλύτερα που μιλάω τώρα και κάνω τώρα τις ερωτήσεις μου, έχοντας ακούσει και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, είναι πιο εύκολο να είμαι πιο συγκεκριμένος σε αυτά που θα πω. Ευχαριστώ κύριε Λάιτινεν για την παρουσία σας και πάλι πάντα είναι πολύ σημαντικό για μας να ακούμε τις ενημερώσεις σας και τις τελευταίες εξελίξεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Frontex. Και πράγματι και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ε, μετατόπιση του κέντρου βάρους. Δεν έχουμε τώρα μεγάλες ροές από την περιοχή του Εύρου στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό έχει να κάνει με τις σημαντικές προσπάθειες και της ελληνικής κυβέρνησης κατά την περίοδο αυτή, αλλά και ε, οφείλονται στη συνεργασία με τη Frontex. Και πάμε τώρα στις ε, ε, διασώσεις στη θάλασσα. Πράγματι έχουμε καλή εμπειρία με τη συνεργασία της Frontex τα προηγούμενα χρόνια. Στον τομέα της εκπαίδευσης, εκατάρτισης κυρίως, καταβάλατε πολύ σημαντικές προσπάθειες για να εκπαιδεύσετε τους δικούς μας εθνικούς ακτοφύλακες. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Τρεις παρατηρήσεις συγκεκριμένα. Πρώτον, είχαμε το μνημόνιο ε, συνεννόησης με τις τουρκικές αρχές που υπογράφτηκε μεταξύ Frontex και Τουρκίας. Και το Μάιο νομίζω. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα η Frontex να είναι και στα σύνορα από την τουρκική πλευρά για να μπορεί να δρά πιο προληπτικά η Frontex ε, σε ό,τι αφορά τη ροή των μεταναστών. Παρόλο που υπογράφτηκε το μνημόνιο αυτό, παρόλο που προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τη συνεργασία μας και να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές, παρόλα αυτά λοιπόν ε, είχαμε ένα πολύ σοβαρό συμβάν επεισόδιο με έναν Τούρκο ακτοφύλακα στις 26 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες ε, πριν. Ε, θα ήθελα τα σχόλιά σας εδώ αν είναι δυνατόν για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Ε, υπήρχε ένα τουρκικό σκάφος της ακτοφυλακής το οποίο ήταν στην, ε, στο, ε, ελληνική, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είχαμε ένα σκάφος από τη Σλοβενία το οποίο ήταν της Frontex, ήταν στη δύναμη της Frontex. Ένα ελληνικό σκάφος πήγε επίσης στην περιοχή. Το τουρκικό ε, σκάφος επικοινώνησε με τα άλλα δύο και είπε ότι έπρεπε να φύγουν. Μετά ε, ενημερώθηκαν ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο γιατί αυτή ήταν η περιοχή της Ελλάδας και μετά συγκρούστηκαν τα δύο σκάφη στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οπότε τι έγινε με τη συνεργασία και το μνημόνιο συνεργασίας. Είστε ικανοποιημένοι ε, μετά το μνημόνιο. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα βγουν θετικά ωφέλη από το μνημόνιο, γιατί εγώ δεν το βλέπω στην πράξη. Δεύτερον, αναφέρατε τα θέματα του προϋπολογισμού. Από ό,τι γνωρίζω, η Κομισιόν πρότεινε να ελευθερώσει 4,5 εκατομμύρια για τη Frontex και για καταστάσεις κατεπίγουσας ανάγκης στην Μεσόγειο. Έγινε αυτό. Ε, το επιβεβαιώνετε. Και είναι αρκετό το ποσό αυτό. Τρίτον, έχουμε την κατάσταση στη Συρία, η οποία μας ανησυχεί πάρα πολύ όλους και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζω και η Frontex να κάνει το ίδιο με τη συνεργασία των εθνικών αρχών των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα τα 4,5 εκατομμύρια ε, αφορούν και τις προετοιμασίες για τυχόν προβλήματα από τη Συρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριος Μούλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα πολλά ενθαρρυντικά. Το πραγματικό πρόβλημα, όπως το είπαν πολλοί ομιλητές mm. ήδη, είναι τι θα γίνει όταν ανακαλυφθεί, εντοπιστεί σκάφος με ανθρώπους στη θάλασσα. Ποια νου ευθύνη είναι μετά, για το τι θα γίνει μετά. Είναι οι εθνικές αρχές, δεν ξέρω αν ε, και υπάρχουν και ενόπλες δυνάμεις που προβλέπονται και ή αν υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο εδώ. Τι κάνουμε, πώς θα συνεργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς οργανισμούς. Και τι προτείνει η Frontex εν προκειμένου. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστα. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις σύντομες ερωτήσεις. Μας είπατε ότι, υπάρχει ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή ακτοφυλακή Δηλαδή, ποιανού αρμοδιότητα θα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πείτε μας περισσότερα για αυτή την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και τι πιστεύουν και τα κράτη-μέλη πάνω σε αυτό. Δεύτερον, ο εξοπλισμός σας. Είπατε ότι πολλά σκάφη δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα με υποδομή, με αυτά που χρειάζονται για τους διασωθέντες. Ε, δεν υπάρχει επαρκής ή καθόλου εξοπλισμό. Για πείτε μας συγκεκριμένα τι σημαίνει πολλά δεν είναι εξοπλισμένα. Το μεγαλύτερο κομμάτι δεν είναι εξοπλισμένο. Ένα κομμάτι και εσείς ως Frontex τι πιστεύετε ότι πρέπει να δαπανίσουμε για αυτούς που σώζονται, για του διασωθέντε ούτω ώστε να κάνουν προτάσεις και συστάσει στα κρατη για το α ή το β. Τρίτο, υπάρχει είδηση και ακούσαμε ότι 1500 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη θάλασσα, πνίγηκαν. Και τι γίνεται με τους ε, νεκρούς, δηλαδή όταν πεθάνει κάποιος και κατά μια επιχείρηση διάσωσης, τι κάνετε αν υπάρξουν θάνατοι. Τέταρτον, η Frontex τώρα έχει μια συμφωνία με το Γραφείο Υποστήριξης θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε και να δούμε το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Λαϊτίνεν για να απαντήσει, ίσως η Κομισιόν θα ήθελε να παρέμβει. Να πει κάτι, σχολιάζοντας τις ερωτήσεις. Λοιπόν, τι έχουμε από την Κομισιόν, ποιος θέλει ίσως να μιλήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις λίγες ερωτήσεις προς την Κομισιόν, αρχίζοντας με το τελευταίο για τη Συρία. Πράγματι, όπως είπαν κάποιοι ευρωβουλευτές, άρχισε μια διαδικασία για την απελευθέρωση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για κατεπίγουσες ανάγκες, όπως είπε και ο κύριος Λάιτινεν, γιατί τον Αύγουστο υπήρξαν ισχυρότατες ενδείξεις ότι θα υπήρχε μια μετατόπιση ε, ε, από τα χερσαία ελληνοτουρκικά προς τα θαλάσσια, εδάφη, ε, θαλάσσια, οδό. στην αρχή ήταν χαμηλά τα επίπεδα από εκεί, γι' αυτό Ε, θεωρήσαμε ότι θα αυξανόντουσαν και θα χρειαζόταν ε, προστασία, υποστήριξη εκεί. Τώρα, το τι κάνει η Κομισιόν και τι προετοιμάζει για να ανταποκριθεί στο συριακό πρόβλημα. Βεβαίως και δουλέψαμε σκληρά πολύ πάνω σε αυτό το θέμα μετά την έναρξη της κρίσης. Αυτό είναι ένα. Τον Αύγουστο μετά από πρωτοβουλία της Κομισιόν δημιουργήσαμε task force ειδικά για τη Συρία. Ε, συνενώσαμε κάποιους οργανισμούς, ε, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Frontex, το ΕΑΖΟ για, τον, για το άσυλο και η Europol, για να δούμε τι γίνεται στην περιοχή και τι μπορούμε να αναμένουμε. Εν τω μεταξύ, Υπήρξαν και αποστολές για να βολιδοσκοπήσουν διερευνητικές, ιδιαίτερα ε, να δουν την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και να δουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Μέχρι τώρα θα έλεγα ότι οι Τούρκοι χειρίζονται την κατάσταση ε, ε, γιατί έχουν ε, φτιάξει καταβλισμούς, αρκετά ικανοποιητικά χειρίζονται την κατάσταση. Υπάρχουν επαφές συνεχιζόμενες εκεί. Βέβαια δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο άμεσο μέλλον. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν παρακολουθούνται εκ του σύνεγγης. Τώρα για το δίκαιο της θάλασσας, κυρία Κέλλερ νομίζω έκανε μια ερώτηση γιατί δεν αλλάζουμε πάλι την εντολή. Ίσως άλλη συνάδελφος ε, δεν μπορεί να απαντήσει, είναι πιο ειδική, αλλά ε, ρώτησε γιατί δεν συμπεριλαμβάνουμε και την έρευνα και τη διάσωση ως καθήκον του οργανισμού. Ακόμα και αν ήταν δυνατόν να υποβληθεί πρόταση της Κομισιόν εδώ, μου φαίνεται ότι δεν είναι μια αρμοδιότητα αυτή που προβλέπουν οι συνθήκες. Οπότε θα ήταν ένα δυσχερέστατο καθήκον αυτό. Ίσως θα έπρεπε πρώτα να μπουν οι διατάξει στη συνθήκη και μετά η Κομισιόν θα είναι υπερευτυχής να ε, υποβάλει προτάσεις με βάση τη συνθήκη. Τώρα όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν. Μου φαίνεται ότι α, απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις που απευθύνονταν στην Κομισιόν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Τώρα λόγο σε εσάς για να κλείσετε, κύριε Λάιτινεν, πριν ε, κάνουμε και κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση για τους συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις που υπέβαλαν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ασχοληθώ με την δυνατότητα αγοράς του εξοπλισμού. Είναι η πρώτη φορά το 2013 δηλαδή όπου εφαρμόζεται η νέα διαδικασία ε, του τροποποιημένου κανονισμού Frontex και όσον αφορά ε, τον ελάχιστο κανονισμό, καθορισμό, συγγνώμη, όσον αφορά τον καθορισμό ελάχιστου εξοπλισμού και όσον αφορά τις ε, συνέργειες. Θα θυμάστε ότι σας είπα ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές στην χρηματοδότηση 100% για το ελάχιστο εξοπλισμό και μέχρι 100% για τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Ακόμα δεν ξέρουμε ε, τι θέληση, ποια είναι η βούληση ε, των κρατών μελών στα πλαίσια της νέας κατάστασης ε, να αναπτύξουν, να χρησιμοποιήσουν τα σκάφη τους. Τον Εύρωτον όταν θα έχουμε τις διμερείς συζητήσεις θα έχουμε καλύτερη ιδέα σύμφωνα με τα μηνύματα που έχουμε από τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της αγοράς ε, του δικού μας εξοπλισμού. Είναι η πρώτη φορά σε αυτό το νέο αλλαγμένο περιφάλλον ε, που σκεφτόμαστε την αγορά του εξοπλισμού. Έχουμε χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες και αυτού του είδους τον εξοπλισμό σε κάποιες επιχειρήσεις. Είχαμε επίσης ε, ανοιχτή ανάπτυξη ε, των ε, ακτεωρών της Ισλανδίας που μας είπαν πάρτε τις και χρησιμοποιήστε τις όπως θέλετε μέσα στα πλαίσια ενός πιλωτικού προγράμματος θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ίδια μέσα. Μια άλλη δυνατότητα είναι η χρήση ε, αγοράς αεροσκαφών ε, για τις ε, εποπτικές πτήσεις. Μέχρι τώρα συνεργαζόμαστε με μια ιδιωτική εταιρεία. Μέχρι τώρα όμως δεν ξέρουμε ακόμα, δεν είμαστε σίγουροι εάν θα κάνουμε προτάσεις αγοράς του εξοπλισμού. Έχουμε αρκετές επιλογές οι οποίες θα ε, εξαρτηθούν από την τελική έκβαση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό. Γιατί σκεφτείτε λίγο ότι και αυτό θα έχει, ο καθαρισμός του προϋπολογισμού θα έχει επίπτωση και σε αυτό. Ε, οι κατευθυντήριες γραμμές, γνωρίζουμε την άποψη του δικαστηρίου για τις κατευθυντήριες ε, γραμμές. Ταυτόχρονα όμως ε, πρέπει να εφαρμόζονται μέχρι ε, να περάσει ο εύθετος χρόνος που χρειαζόμαστε, ο εύλογος χρόνος ε, για να υπάρξουν οι απαραίτητες αλλαγές. Ακόμα βασίζονται οι θαλάσσιες επιχειρήσεις στις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες τώρα έχουν καταργηθεί. Δεν έχουμε ασχοληθεί. Δεν έχουμε βρεθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι σε ε, ε, εντατική βάση ε, για να συζητήσουμε την αλλαγή των κατευθυντηρίων γραμμών. Μην ξεχνούμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ δύσκολης συζήτησης. Για την ερώτηση κυρία Σκέλλερ, νομίζω ότι να πω το εξή. Εγώ προσπαθώ να ρίξω μια αναδρομική ματιά στις διαδικασίες. Κανεί δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Θα πρέπει να έχουμε κάποια βάση όμως για να σχεδιάσουμε τις ε, δραστηριότητε μας. Και αυτό ε, που ήθελα να πω είναι ότι ε, οι περιπτώσεις έρευνας και διάσωση στη θάλασσα δεν είναι η εξαίρεση. Είναι κανόνα στις επιχειρήσεις μας. Ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει να καθορίσουμε δύο διαφορετικά σκέλη αυτής της ε, θαλάσσιας διάσωσης. Εάν συζητήσουμε με δικηγόρους, ε, τότε θα ξεκινήσουν ατέρμονες συζητήσεις σχετικά με το τι προβλέπει ε, η διεθνής νομοθεσία κτλ. Το ξέρουμε αυτό. Εγώ ε, ε, είμαι ε, αυτός ο οποίος ασχολείται με την πρακτική πλευρά του, την πρακτική πλευρά του θέματος. Δεν με ενδιαφέρει αν η νομοθεσία η οποία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσω είναι διεθνής ή ενωσιακή πώς προωθήσαμε τι δραστηριότητε μα όσον αφορά τι δραστηριότητε, έρευνα και ε, διάσωση, εμεί θελήσαμε να είμαστε πάντα ε, έτοιμοι, να έχουμε πάντα σε ετοιμότητα ένα κέντρο, ε, να γνωρίζουμε ανα πάσα στιγμή που βρίσκονται και ποια είναι τα μέσα τα οποία μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας, πόσο γρήγορα μπορούμε να τα αναπτύξουμε και να φτάσουν επί τόπου και αυτήν την ικανότητα θέλουμε να βελτιώσουμε. Γιατί ε, όταν μια τέτοια κατάσταση ε, προκύψει, το κέντρο θαλάσσιου συντονισμού, θαλάσσιου επιχειρησιακού συντονισμού αναλαμβάνει ε, όλο το βάρος της ανάπτυξης ε, των, ε, του εξοπλισμού και των μέσων που έχουμε στην διάθεσή μας και βεβαίως εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε η ταυτοποίηση, δηλαδή ε, ε, στο, το, ε, ότι να υπάρχει ένας μονάχα υπεύθυνος οργανισμός με τον οποίο θα συνεργαζόμαστε. Τρίτον, στην κεντρική Μεσόγειο και κυρίως από, την από τον Οκτώβριο και μετά ξεκινάει μία περίοδος ήπιων καιρικών συνθήκων και γι' αυτό ακριβώς τότε έχουμε αύξηση των ε, λαθρομεταναστών. Το είδαμε και πέρσι, το είδαμε ε, και σε άλλες ε, περιπτώσεις και προσαρμοζόμαστε και εμείς σε αυτόν τον ρυθμό που οδηγούνται οι διασωθέντες μετανάστες. Αυτό το αποφασίζει η αρμόδια Εθνική Αρχή. Το 2011 περίπου 60.000 διασωθέντες βρέθηκαν ε, ε, σε ιταλικά ε, ύδατα υπό την, υπό τον συντονισμό των Ιταλικών συντονιστικών αρχών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγήθηκα στη Λαμπεντούζα. Δεν γνωρίζομαι ακριβώς ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί γιατί ξεπερνάει τον έλεγχο των συνόρων. Αυτό όμως μαθαίνουμε και αυτό κατεγράφει η ακτοφυλακή είναι σημαντική εμπλεκόμενη φορείς. Οι κύριοι εμπλεκόμενοι λοιπόν και οι κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι η ε, Τα θέματα του προϋπολογισμού. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τις ε, τροπολογίες, τις τροποποιήσεις μάλλον του προπολογισμού 2013. Ε, όλα αυτά τα οποία σχετίζονται και με τα θέματα Σέγγεν ε, μιλούμε τώρα για αυτές τις αβεβαιότητες τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και οι οποίες δεν μας επιτρέπουν τον σωστό και ομαλό προγραμματισμό.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 ξέρουμε πάρα πολύ καλά ε, και τις εμπειρίες του παρελθόντος. Ξέρουμε ότι όταν ας πούμε συνέβη, ε, ε, αναφέρομαι στην Συρία, ξέρουμε ότι όταν συνέβησαν τα συμβάντα της Λιβύης υπήρχαν τμήματα της Μεσογείου τα οποία ορίστηκαν ως εμπόλεμες ζώνες και στις οποίες δεν μπορούσαμε πλέον να έχουμε δυνατότητα επιχειρησιακής παρέμβασης. Ε, το θέμα της Frontex ε, σχετικά με την, ε, με την τουρκική ακτεωρό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ε, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά τις ε, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πρώτον, ο καθένας έχει υποχρέωση που είναι παρόν, δηλαδή ε, στην περιοχή, να δώσει βοήθεια. Ασχέτως αν είναι ιδιώτης, πλειοκτήτης, αν είναι απλό σκάφος, στρατιωτικό σκάφος, από τη στιγμή που υπάρχει μια κλίση από το κέντρο συντονισμού, πρέπει κανείς να συμμετάσχει εφόσον βρίσκεται στην περιοχή. Η δεύτερη, το δεύτερο σημείο που ήταν ε, η περίπτωση, στην περίπτωση που αναφέρατε, οι τουρκικές αρχές ε, ήταν ε, υπεύθυνε για το επεισόδιο το οποίο έλαβε χώρα 15 μίλια από την τουρκική, 15 μέτρα από την τουρκική ακτή το κέντρο, το κέντρο ε, ε, από την τουρκική πλευρά ήταν ε, αυτοί οι οποίοι έπρεπε να παρέμβουν. Έγινε μία προσφορά, δεν δέχτηκαν όμως να πάρουν τη βοήθεια αυτή. Όσον αφορά το αποθεματικό των 4,2 εκατομμυρίων, κύρια αιτιολόγηση είναι ότι ε, είδαμε ε, να μετατίθεται πάρα πολύ γρήγορα το κέντρο βάρους από τα χερσαία σύνορα στα θαλάσσια ε, και αυτή η, και, και μάλιστα επικέντρωση μεγάλη στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολλά εναέρια μέσα, ε, χρησιμοποιούνται σκάφη ταχείας ε, επέμβασης κτλ. Ε, κοντεύουμε στο τέλος του χρόνου, 86% έχουν, των κονδυλίων έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, επομένως θέλουμε επιπλέον χρήματα, επιπλέον κονδύλια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις νέες επίγουσες ανάγκες και ένα τμήμα της δικαιολόγηση για τα, αυτά τα 4,5 διορθώνω, 4,5 ε, εκατομμύρια είναι βεβαίως και η κατάσταση στην Συρία, διότι υπάρχει σαφής διασύνδεσης ανάμεσα ε, σε αυτά τα δύο θέματα. Τέλος, το ζήτημα για την ακτοφυλακή. Αναφέρθηκα στη λειτουργία της ακτοφυλακής εγώ αναφέρομαι στην, ε, στην λειτουργία, στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Σε αυτήν την ε, περιοχή συμμετέχει η Ακτοφυλακή και οπωσδήποτε εμείς δεν θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε ένα υπερεθνικό σώμα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει σωστός συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και όλων των εμπλεκομένων. Υπήρξε ένα ερώτημα σχετικά ε, σχετικά με το κατά πόσον ε, είναι καλά ή όχι καλά εξοπλισμένα τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Η απάντηση είναι ότι ο εξοπλισμός των ε, σκαφών είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε μία checklist που βλέπουμε ότι όλα έχουν γίνει σωστά, ότι υπάρχει ένα πακέτο τυποποιημένο το οποίο καλύπτει τις βασικές ανάγκες των περιοχών γιατί υπάρχουν ας πούμε κάποιες ε, περιοχές ε, οι οποίες ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες όπως η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος ας πούμε. Ελπίζω ότι απάντησα στα κυριότερα ερωτήματά σας. Ε, είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως για περαιτέρω ερωτήματα ε, και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε μου δώσατε τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαϊτίνεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια την οποία καταβάλατε έτσι ώστε να απαντήσετε. αλλά και η κυρία Κέλλερ και ο κύριος Τριανταφυλλίδης θέλουν ε, να αντιδράσουν ή να ε, θέσουν να υποβάλουν ένα επιπλέον ερώτημα και ο κύριος ε, Παπα-Νικολάου βλέπω. Η κυρία Κέλλερ πρώτα. Και μετά εσείς κύριε Τριανταφυλλίδη. Um, Ευχαριστώ πολύ. Δύο σύντομες συμπληρωματικές. Λέτε ότι η τροπολογία είναι για έγινε για τον προπολογισμό του 2013, γιατί εμεί πήραμε τον προπολογισμό για το 2012. Πήραμε λάθο τροπολογία. Δηλαδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φέτο τα χρήματα πια, οπότε είναι άκυρη η ε, τροπολογία. Δεν το κατάλαβα. Για ποιο χρόνο θέλατε τα πιο πολλά χρήματα. Επίση, για το ίδιο θέμα. Λέτε ότι χρειάζεστε περισσότερα χρήματα γιατί υπάρχει αυτή η μετάβαση από τα χερσαία στα θαλάσσια σύνορα. Αλλά ναι, έλεγα ότι τώρα είναι αποκλεισμένα τα χερσαία, δεν μπορούν να περάσουν από τα χερσαία. Ε, αυτό έλεγα κι εγώ. Οπότε τώρα χρησιμοποιούνται χρήματα για να κλείσουν τα χερσαία, μετά πάνε στη, στα θαλάσσια και μετά θέλετε χρήματα για να κλείσετε και τα θαλάσσια. Ε? Μάλιστα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν μου απαντήσατε για το αν γίνονται αναχαιτήσεις στη θάλασσα και για, το, για τη Συμφωνία Συνεργασίας Frontex-EASO. Κύριε Μούλτερ, θέλετε κι εσείς. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Ποια είναι η, σε τελευταία ανάλυση, ποια είναι η ευθύνη, ποια είναι η ε, ε, ευθύνη, αν δηλαδή ε, διασωθούν κάποιοι, χαιρετιστούν κάποιοι, τι θα γίνει μετά, ποια είναι η μοίρα τους. Ο κύριο Πάπα Νικολάου, κύριε Λάιτινεν, νομίζω υπάρχει μια παρεξήγηση. Εγώ αναφέρθηκα σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου. Όχι στις 6, ίσως αναφέρεστε σε ένα συμβάν όπου έγινε προσπάθεια διάδοσης 50 μέτρα από την τουρκική ακτοφυλακή και χάθηκαν ζωές τότε. Δεν λέω αυτό. Λέω για μία σύγκρουση μεταξύ ενός περίπου ενός, ε, μιας ακτορού ε, και του σλοβενικού σκάφους και της Frontex. Πολύ σύντομα. Frontex εάζω και εργασία συμφωνίας. Δεν μας είπατε τίποτα γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Λάιτινεν, ε, σας δίδεται δεύτερη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχω πάνω από ένα δευτερόλεπτο για τη δεύτερη ευκαιρία. Τώρα, οι τροπολογίες για τον προϋπολογισμό. Μιλάω για το 2013, δηλαδή τις πρώτες ψηφοφορίες. Υπάρχουν δύο αποθεματικά που ψηφίζουμε. Το ένα είναι τα 4,5 που μιλάμε και το άλλο ήταν το 75% των επιχειρησιακών ε, ε, δαπανών όλου του οργανισμού ε, λόγω του Σέγγεν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι σημαίνει για τον οργανισμό η αυτή η αβεβαιότητα αν θα πάρουμε το 25% των επιχειρησιακών δαπανών. Ή το 100%. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια ότι δηλαδή απορρίφθηκαν, καλά νέα, απορρίφθηκαν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών οι σχετικές τροπολογίες. Ωραία. Τώρα για τις αναχαιτήσεις στη θάλασσα. Όπως ξέρετε, κανενός είδους αναχαιτήσεις δεν γίνονται στη θάλασσα εκτός αν πρόκειται για διάσωση και συνοδεία μέχρι σε ένα ασφαλές σημείο αποβίβασης. Ε, αυτά είναι από παλιά. Τώρα δεν γίνονται αποθήσεις τόσο πολύ. Είναι σαφές ότι ε, αναφέρεται ρητά στις επιχειρήσεις που μετέχει η Frontex ότι δεν μπορεί να γίνει απόθεση. Να παγυρίσουν πίσω. Τώρα, ποια, ποια είναι η ε, ευθύνη σε τελευταία ανάλυση. Ε, ελπίζω να μην έδωσα, προσπάθησα να μην δώσω την εντύπωση ότι πάω να ξεφύγω από τις ε, ευθύνε μας. Γι' αυτό είπα ότι ε, οι νομικοί έχουν τις απόψεις τους, αλλά και οι πρακτικοί τις δικές τους. Ε, πάντοτε θα πρέπει να αποφασίζει η αρμόδια εθνική αρχή. Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο των συνόρων και τις κοινέ επιχειρήσεις γιατί η χώρα υποδοχής έχει το, τη γενική διοίκηση και το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις θαλάσσιας ε, έρευνας και διάσωσης. Η ευθύνη πιστεύουμε ότι είναι να προαγάγουμε τις βέλτιστες πρακτικές και την καλή έκβαση αυτών των επιχειρήσεων όσο περισσότερο μπορούμε. Τώρα, το η περίπτωση της 26ης Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω τη λεπτομερή έκθεση, αλλά ξέρουμε ότι ήταν μια περίπτωση όπου ένα σκάφος που συμμετείχε στις ε, συντονισμένες επιχειρήσεις της Frontex υπό τη διοίκηση της ακτοφυλακής συνεκρούστη με μια, ε, ένα σκάφος τουρκικής ακτοφυλακής σε μια περίπτωση όπου υπήρχε αμφιβολία σχετικά με τη θέση του σκάφους, αν ήταν, σε ποια χωρικά ύδατα ήταν. Ε, τώρα, συνεργασία Frontex-EASO. Ε, είμαστε πολύ ευτυχείς και μάλιστα ήμουν ε, παρόν πριν από ένα μήνα στη ε, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου, Συμβουλίου Διαχείρισης και ένα συνάδελφος ήταν και στην άλλη συνεδρία 26 Σεπτεμβρίου και τότε υπογράφηκε και η συνεργασία μεταξύ Frontex και Άζο. Δεν αρχίσαμε από το μηδέν, ε, ε, έχει προηγηθεί συνεργασία μέχρι τώρα γιατί η Frontex βοήθησε την Άζο να αντιμετωπίσει τις διαδικασίες και τα διοικητικά. Κάναμε πολύ κοινή δουλειά για την ανάλυση του κινδύνου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων, την αύξηση ε, των μέτρων ε, και των ικανοτήτων και ξέρουμε πώς θα αναπτυχθεί η συνεργασία με ανταλλαγή πληροφοριών, επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση και βελτίωση της ε, ποιότητας του screening. Εκεί δουλεύουμε πάρα πολύ. Ε, πρώτη εξέταση. Η ΕΑΖΟ είναι πιο έμπειρη ε, σε θέματα που αφορούν τη χώρα προέλευσης, ενώ εμείς γνωρίζουμε καλύτερα τους διάφορους κανόνες ε, που διέπουν τη διέλευση των συνόρων. Μόλις μπορέσουμε να συγχωνεύσουμε τις πληροφορίες μας, τότε οι εμπλεκόμενοι θα έχουν καλύτερη εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία. Μίλησα ήδη για το screening, που είναι, αν θέλετε, ε, μια πρώτη εξέταση για να δούμε αν οι ε, μετανάστες θα πάνε σε διαδικασία ασύλου ή αν αυτό δεν συμβαίνει θα ακολουθήσουν άλλες διαδικασίες. Και ενδεχομένως αν τελευταία ε, ναι, να ξαναγυρίσουν σε, ή διαδικασία, να μπουν σε διαδικασίες επιστροφής. Ευχαριστούμε κύριε Λάιτινεν, εκτιμούμε την προσπάθειά σας να αντιμετωπίσετε ε, τα, τις ανησυχίες των μελών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Λοιπόν, σταματούμε εδώ αυτή μας την ε, επαφή. Την περασμένη εβδομάδα έγινε δεκτή τροπολογία για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Frontex, αυτού του οργανισμού. Ε, θα χαρούμε να σας ξαναδούμε σύντομα και σε λίγα λεπτά θα αρχίσει και κλεισμένον των θυρών η συνεδρίαση των συντονιστών. Όσοι δεν θα συμμετάσχετε, δεν έχετε δουλειά στην συνεδρίαση των συντονιστών, παρακαλώ να εγκαταλείψετε σιωπηλά την αίθουσα.